Um, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε. Κοινή συζήτηση για την τελευταία έκθεση πρόοδου για την εφαρμογή της, ε, του θεματολογίου της Ένωσης για τη μετανάστευση και δύο νέες νομοθετικές προτάσεις. Μία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για τους ε, Ευρωπαίους ε, συνδέσμους και την άλλη για τις θετικές για την μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Δεν ξέρω αν οι διερμηνείς θέλουν να κάνουν μια δήλωση. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, η έκθεση προόδου θα ασχοληθεί με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, την κατάσταση όσον αφορά τις μεταναστευτικές οδούς και την ανάγκη να βελτιωθούν οι ε, ρυθμοί των επιστροφών και για τη δήλωση μεταξύ ε, Ευρώπης και Τουρκίας που έχει συζητηθεί. Τονίζει τη σημασία και του μεταρρυθμισμένου Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου και θέλει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση όπως πρότεινε ήδη η ΛΥΜΠΕ μέσω της έκθεσης Μετσόλα και Έγκε του 2016 μια ολιστική αντιμετώπιση για τη μετανάστευση. Μία από τις πρωτοβουλίες που υπέβαλε η έκθεση μέσω αυτής της ε, έκθεσης είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια συντονισμού με τους βασικούς εταίρους μας στις ε, σημαντικές τρίτες χώρες. Και εδώ έχουμε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τους ε, συνδέσμους μετανάστευσης που η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη αποστέλουν στις ε, μη κοινωνικέ χώρες. Επίσης, χρειαζόμαστε καλύτερες στατιστικές για την πολιτική μας για το άσυλο και τη μετανάστευση και, αυτό επιδιώκει, και αυτό επιδιώκει να επιτύχει η Eurostat με την πρόταση για την τροποποίηση του ενισχύ κανονισμού για τις στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Πρόσταση αυτή συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση αποτελέσματα για το θεματολόγιο της Ένωσης στην μετανάστευση που παρουσίασε στην Επιτροπή μας ο Επίτροπος Αβραμόπουλος τον περασμένο Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτεμβρίου. Πρώτα έχουμε τρει ομιλητές πριν έχουμε συζήτηση. Πρώτα απ' όλα την κυρία Μάρτα Σίγκαν που είναι διευθύντρια για τη στρατηγική και τι ε, γενικέ υποθέσει στην Γενική Διεύθυνση Home. Θα μα παρουσιάσετε κύριε σημεία που σχετίζονται με την πρόοδο στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θυματολογίου για την Μετανάστευση. Μετά θα έχουμε την κυρία Σιμώνα Αρντοβίνο, που είναι υπάλληλο ε, στην ε, μονάδα για την παράτιμη μετανάστευση και την πολιτική επιστροφών για 7 λεπτά και τέλος θα έχουμε τον κύριο Βρόνσκι, τμήματάρχη στο Eurostat για 7 λεπτά. Πρώτα λοιπόν να δώσω λόγο στην κυρία Σίγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Όπως είπατε, η Επιτροπή 16 Μαΐου ενέκρινε το, την έκθεση πρόοδου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση. Και θα σας παρουσιάσω λοιπόν ε, την πρόοδο που επετεύχθη κατόπιν της εκθέσεως του Μαρτίου. Είναι η τρίτη έκθεση που καλύπτει τις ενέργειες που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και εντοπίζει τις συγκεκριμένες δράσεις που είναι βασικές για την αποτελεσματική αντίδραση της Ένωσης στη μετανάστευση. Η έκθεση καταδεικνύει ότι η κατάσταση για τις κύριες μεταναστευτικές διαδρομές έχει περαιτέρω σταθεροποιηθεί στην περίοδο αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο από ένα υψηλό τον Οκτώβριο του 2015 10.000 των ε, αφήξεων ε, ανά ημέρα. Μετά την εφαρμογή της δήλωσης με την Ένωση και την Τουρκία έχουμε μεγάλη ε, πτώση. Επίσης στην ε, Κεντρική Μεσόγειο και μετά την ε, συνεργασία μας με την Ιταλία, την ε, Λιβύη, την Ιζέρ και άλλες ποσαχάριες χώρες οι αφήξεις έχουν μειωθεί κατά 81% το 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Για την Δυτική Μεσόγειο, εδώ έχουμε αύξηση των αφήξεων, αλλά ήταν χαμηλή η βάση και αναλαμβάνεται δράση για να ελεγχθεί η κατάσταση. Ο συνολικός αριθμός αφήξεων στην Δυτική Μεσόγειο είναι 17.320. 82% περισσότεροι από την αντίστοιχη περίοδο του 17. Νομίζω ότι αξιόλογο είναι να αναφέρω, όπως και η έκθεση, για την διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων. Η κατάσταση παραμένει σταθερή αλλά μια υποδιαδρομή μέσω Ελλάδα, Αλβανία και Βοσνία Αζεγοβίνης στην Κροατία και άλλε χώρε εκεί έχει αυξηθεί λοιπόν η κίνηση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση μέσω τακτικών βίντεο συσκέψεων. Η αύξηση των αφήξεων σημαίνει ότι έχουμε και λιγότερους πνιγμούς και η πρόληψη αυτών των πνιγμών που εξακολουθούν δυστυχώς πολύ συχνά να συμβαίνουν πάνω από 1412 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, φέτος. Αυτό θα εξακολουθήσει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Επίσης έχουμε πολύ αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε 1222 υπαλλήλους που βοηθούν ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Συνοροφυλακής και Ακτοφυλακής που βοηθούν την επιτήρηση των συνόρων στη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Και επίσης έχουμε και μία εφεδρεία 400-500 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν υπάρχουν προβλήματα. Περισσότερη πρόοδος επετεύθη όσον αφορά την χρηματοδοτική και λειτουργική στήριξη στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν έντονη μεταναστευτική πίεση. Ιδιαίτερα τα κράτη που ασχολούνται κυρίως με τα θέματα αυτά στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Ισπανία. Επίσης έχουμε περίπου διπλασιάσει την προσπάθεια και οικονομικά 22 δις μεταξύ 15 και 18 σε σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη 9,6 δις. Τα hotspot λειτουργούν σωστά, ούτως ώστε όλοι οι αφιχθέντες να καταγραφούν και να πάρουμε τα δακτυλικά τους ε, αποτυπώματα. Η συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή η Europol και η υπηρεσία ασύλου έχουν λάβει περισσότερους πόρους και χρησιμοποιούν επιτόπου εμπειρογνώμονες. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής στα hotspot και για να αυξηθούν οι εθελούσιες επιστροφές. Η έκθεση επίσης αναφέρει ότι ενισχύσαμε τις σχέσεις με τις χώρες προέλευσης και μετάβασης μέσω ενός αποτελεσματικού πλαισίου μέτρων για να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση, να βοηθήσουμε τους ε, γνήσιους πρόσφυγες και να βοηθήσουμε την ε, ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Αναφέρουμε στην εφαρμογή της δήλωσης Ελλάδας και Τουρκίας, που είναι επίσης κάτι που εντάσσεται και στο πλαίσιο συνεργασία που έχουμε για τις σχέσεις με την Αφρική και ιδιαίτερα για την ε, Βόρεια Αφρική και τη συνεργασία με τις χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Μεταξύ τη έγκρισης και τη έκθεση ε, και του σήμερα έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε τονίζω ότι εντωμεταξύ ένα από τα απτά άμεσα αποτελέσματα ήταν η συμφωνία να περάσει από το αποθεματικό του Ταμείου Ανάπτυξη ε, μισό δισεκατομμύριο στο καταπίστευμα για την Αφρική. Η Επιτροπή έχει ήδη προετοιμάσει την απόφαση για να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση. Θα την υποβάλουμε στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη τον Ιούλιο. Επίσης, επευκαιρία. Τονίζω ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει πάντα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στα καταπιστεύματα γιατί χρειαζόμαστε ακόμα μισό δισεκατομμύριο για αυτό το καταπίστευμα συγκεκριμένα για την Αφρική. Περαιτέρω. Ελπίζουμε σύμφωνα να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τη χρηματοδότηση του δεύτερου τμήματος της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Αναφερθήκατε στα προγράμματα επανεισδοχής και επανεκατάστασης. Η επανεκατάσταση έχει μειώσει την πίεση για τα κράτη πρώτης γραμμής και έχουμε δώσει βοήθεια σε πολλά άτομα που προσπαθούν να διαφύγουν από κινδύνους. Έχουμε δύο προγράμματα επανεκατάστασης που βοήθησαν 32.000 από τα πιο βάλατα άτομα να καταφύγουν στην Ένωση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα επανεγκατάστασης 50.000. Τα κράτη-μέλη έκαναν ε, τη μεγαλύτερη ομαδική δέσμευση που έχει γίνει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι αφαιρέσαμε από τα απάνθρωπα κυκλώματα διακινητών τα θύματα τους και δίνουμε ασφαλή ε, πρόσβαση στα άτομα που τη δικαιούνται. Αυτό καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα γίνει φρούριο. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας να παίζουμε υπεύθυνο ρόλο και να δίνουμε προστασία σε αυτούς που τη χρειάζονται. Η επανεκατάσταση πρέπει να γίνει το μόνιμο μέλλον της ε, κοινή πολιτικής μας για το άσυλο. Αλλά όπως κατέδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα, δεν εφησυχάζουμε. Πολλές ζωές χάνονται στη θάλασσα και πριν φτάσουν καν στη θάλασσα. Θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε τις τάσεις για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση και για να έχουμε μια βάση για την ε, πολιτική μας. Γι' αυτό είναι ουσιώδες να συνεχιστούν οι τακτικές εκθέσεις που υποβάλλουμε και να επαγρυπνούμε για τι νέε διαδρομέ που μπορεί να προκύπτουν από τον ε, Μάιο. όπω είπα πολλά συνέβησαν ιδιαίτερα οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ασχολήθηκε πολύ με τη μετανάστευση και τα πορίσματά του επαναβεβαιώνουν την ολιστική μας προσέγγιση για τη μετανάστευση που συνδυάζει πιο αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, αυξημένη εξωτερική δράση και τις εσωτερικές πλευρές με βάση και τις αρχές και αξίες μας. Οι ηγέτε βοήθησαν να δοθούν πόροι για να αντιμετωπιστούν ε, τα βασικά αίτια της μετανάστευσης και στήριξαν την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νέα πρόταση για να αυξηθούν οι επιστροφές και για να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου στα εξωτερικά σύνορα. Επίσης συμφώνησαν να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ασύλου όσο ταχύτερα γίνεται και να προωθηθεί και η περιφερειακή συνεργασία για την αποβίβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τις βασικές δράσεις όπως τις εντοπίσαμε στην έκθεση πρόοδου του Μαΐου. Ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα αφορά τις συμφωνίες για συνεργασία μεταξύ της ε, δική μα ε, συνοριακή και εκτοφυλακή και τι αντίστοιχε υπηρεσίε των Δυτικών Βαλκανίων και επίση δίνουμε λειτουργική βοήθεια στι υπηρεσίε αυτέ αυτών των χωρών. Για παράδειγμα, στην Αλβανία. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει μια απόφαση για την υπογραφή αυτή τη συμφωνία την τρέχουσα εβδομάδα. Και για την ε, Φύρομ συμφωνήσαμε τον Απρίλιο και για το Μαυροβούνιο έχουν ε, μόλις εκκινήσει οι διαπραγματεύσεις και επίσης θα δοθεί επίγουσα βοήθεια προς τις Ιταλικές αρχές. Είναι σε φάση ολοκλήρωση η διαδικασία και οι προσπάθειες ε, της ΥΠΑ ε, της Αρμοστίας των ΗΠΑ σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη συνεχίζουν τα προγράμματα του επιγόντος μηχανισμού μεταβίβασης. Από τη Λιβύη έφυγαν 158 άτομα και 1378 επανεκαταστάθησαν μετά από αιτήματα 1987. Συνεχίζουμε τη μετακατάσταση. Πολύ λίγα άτομα πρέπει να μετακατασταθούν από την Ιταλία. Ο συνολικός αριθμός των ε, μετα... Ε, μεταεγκαταστηθέντων είναι 400, 600, 4.600 περίπου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμεθα μεταξύ των διαφόρων εκθέσεων πρόοδου και θα συνεχίσουμε και περαιτέρω. Η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα πήρε σημαντικές αποφάσεις. Αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε το πρώτο άτυπο συμβούλιο υπό την Αυστριακή Προεδρία. Συνεχίζεται λοιπόν η δουλειά και στηριζόμεθα και σε εσά για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρντουβίνο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της αναδιατύπωσης ε, της ε, υφιστάμενης νομοθεσίας 3774 ε, του 2004 όσον αφορά τους Ευρωπαίους αξιωματούχους σύνδεσης μετανάστευσης που προβλέπει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το ρόλο των κρατών μελών και των αξιωματικών σύνδεσης που θα μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες όπως επίσης και για τη δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης των αξιωματικών αυτών σύνδεσης μετανάστευσης στις τρίτες ε, χώρες. Κατά το 2016 με 2017 κάναμε μια διεξοδική αξιολόγηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που έδωσε τη δυνατότητα της πρώτης αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας και που έδισε επίσης ε, τα στοιχεία, ε, τα αποδεικτικά που χρειάζονταν για την αναδιατύπωση αυτή με την, ε, τα πορίσματα της αξιολόγησης αυτής ε, καταλήξαμε σε δύο συμπεράσματα. Καταρχά, οι 500 εξωματικοί σύνδεσης περίπου που αναπτύσσονται σε τρίτες χώρες από τα κράτη-μέλη, που στέλνονται σε τρίτες χώρε από τα κράτη-μέλη, είναι πολύτιμες, ε, πολύτιμα ε, στοιχεία που μας επιτρέπουν να, διαχειριστούμε τις ε, μεταναστευτικές πιέσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλήρε δυναμικό των συνδέσμων αυτών, των αξιωματικών σύνδεσης ε, και δεν ήταν επαρκές το δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των αξιωματούχων αυτών προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. Ε, η, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ε, ε, έρθει σε επαφή μαζί τους, έχουμε συνεργαστεί μαζί τους και στις Βρυξέλλες και μέσω εργαστηρίων ε, συνδρομής σε όλο τον κόσμο όπου δραστηριοποιούνται και καταλήξαμε ε, ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητα και τις υποδομές που παρέχουμε στους αξιωματούχους και να τα καταγράψουμε σε ένα νέο κείμενο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη και πρόσφαση, πρόσφατη ε, τάση ε, αποστολή των αξιωματούχων αυτών στις τρίτες ε, χώρες. Στις 16 Μαΐου λοιπόν η νομοθεσία που δημοσιεύθηκε προσπαθεί να ε, δημιουργήσει ένα, ένα δίκτυο ε, στο πλαίσιο του οποίου θα δια, δραστηριοποιούνται οι αξιωματούχοι αυτοί. Ε, δεν είναι νέα βέβαια η ιδέα. Προσπαθήσαμε να βασιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στην υφιστάμενη νομοθεσία γιατί πρόκειται για αναδιατύπωση, δεν είναι νέα πρόταση και θα δείτε στα καθήκοντα των ανθρώπων αυτών τις κοινέ μας προσδοκίες όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, μια ισχυρή συνεργασία κατά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, όπως επίσης και της πρόληψης εγκληματικής δραστηριότητας, όπως της ε, λαθρεμπορίας μεταναστών όπως επίσης για το θέμα των ε, εισδοχών ε, από τις τρίτες χώρες ε, και ο σημαντικός ρόλος βέβαια των ανθρώπων αυτών όσον αφορά τα προγράμματα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Κάτι πολύ σημαντικό είναι επίσης η συνεργασία των αξιωματούχων αυτών επιτόπου. Λάβαμε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση των αξιωματούχων σύνδεσης μετανάστευση. Προτείνουμε λοιπόν λοιπόν να υπάρξει μία, ένα συμβούλιο διαχείρισης ε, το οποίο θα διαχειρίζεται την ε, υποστήριξη αυτών των ανθρώπων και ο στόχος είναι το Συμβούλιο αυτό να είναι ένα δυναμικό σώμα που θα δίνει μια καθοδήγηση μακροχρόνια επιτόπου στους αξιωματήχους, αλλά και ε, ενημέρωση για πρακτικά ζητήματα καθημερινά, τα οποία θα είναι κοινού ενδιαφέροντος. Επομένως, έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο ε, ζωντανό τρόπο αντιμετώπισης ε, των προβλημάτων. Επίση προσπαθούμε να καλύψουμε, να προβλέψουμε τις ε, αναδυόμενε τάσει ε, και να δούμε πώς μπορούν να δραστηριοποιούνται και να αποστέλλονται οι αξιωματούχοι σε περιοχές, σε διαδρομές που προκύπτουν, που αλλάζουν συνεχώς. Η επαφή με τι τοπικέ με είναι επίση πάρα πολύ σημαντική και προσπαθούμε επίσης να γνωρίσουμε κοινού ε, στόχους. Υπάρχει επίσης και μία πρόκληση όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας ε, των εθνικών αξιωματούχων και ε, για να μην υπάρξει αναστάτωση του τρόπου με τον οποίο εργάζονται αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε αυτά τα στοιχεία του, της νομοθεσίας που είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικά και που δεν έχουν πάρα πολύ επιχειρησιακή αξία, όπως για παράδειγμα η ε, υποβολή εκθέσεων σε διετή βάση. Όσον αφορά την επεξεργασία τώρα των ε, ε, προσωπικών στοιχείων ε, των αξιωματούχων και τη δραστηριοποίηση του σε τρίτε χώρες, πρέπει να υπάρχει απαραίτητη νομική κάλυψη, κάτι το οποίο κάνει η καινούρια νομοθεσία και αφορά βέβαια τα προσωπικά στοιχεία που θα, θα επεξεργάζονται οι αξιωματούχοι αυτοί κατά την διεκπαιρέωση των καθηκόντων τους για την επανεγκατάσταση και τις διαδικασίες εισδοχής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το ε, Συμβούλιο αυτό διαχείρισης ε, ε, και πώς θα αναφέρεται αυτό στο διετές επιχειρησιακό πλαίσιο. Υπάρχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα μικρής κλίμακας, μελέτες, ε, αναλυτικά προγράμματα, κατάρτιση, εκδηλώσεις, εργαστήρια, σεμινάρια για τους ε, ε, αξιωματούχους και οι ίδιοι μπορούν μάλιστα να κάνουν να οργανώνουν τέτοιου είδους σεμινάρια με τις δεξιότητες που θα έχουν. Εμείς με χαρά περιμένουμε να συνεργαστούμε με εσάς, με τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να ολοκληρώσουμε αυτήν την νομοθεσία. Κύριε Βρόνσκι, 7 λεπτά. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα παρουσιάσουμε την τροπολογία του κανονισμού 2007 για την μετανάστευση και την διεθνή προστασία. Η παρουσίαση θα γίνει από τον συνάδελφό μου. Η κυρία Σίγκαν που μίλησε προηγουμένως χρησιμοποίησε πολλά στατιστικά στοιχεία, πολλά δεδομένα. Μας έδωσε ένα παράδειγμα για τα στοιχεία της Eurostat που βοηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών. Κάποια από τα στοιχεία αυτά μπορεί να έρχονται από τη βάση δεδομένων της Eurostat. Απλούστατα γιατί η συλλογή δεδομένων της Eurostat δεν είναι ενημερωμένη Γι' αυτό και τα στοιχεία που χρησιμοποίησε δεν ήταν αποκλειστικά από τη Eurostat. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη συλλογής πιο ολοκληρωμένων, πιο ενημερωμένων, πιο συχνών στατιστικών στο πεδίο αυτό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που προκύπτει από την αυξημένη είσοδο υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης της μετανάστευση, αλλά και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στατιστικές στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευση, καλύπτονται από στατιστικά για το άσυλο αλλά και Επίση στον τομέα εφαρμογή τη νομοθεσία σχετικά με την μετανάστευση. Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται στους υπάρχοντες κανονισμούς 622 του 2007. Επιπλέον χρησιμοποιούμε τον κανονισμό της Επιτροπής 216 του 2010. Υπάρχουν και άλλες νομικές πράξεις που είναι σχετικές, για παράδειγμα η οδηγία για τις άδειε παραμονές, αλλά και άλλες οδηγίες. Η Eurostat συλλέγει δεδομένα βασιζόμενη σε αυτές τις οδηγίες και άλλες νομικές πράξεις. Επί του παρόντος όμως οι στατιστικές ανάγκες μπορούν να βοηθηθούν από την εθελοντική συλλογή δεδομένων, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Από 20 μέχρι 28 χώρες προσφέρουν δεδομένα, αλλά δεν έχουμε τρόπο να τα ελέγξουμε. Η έκθεση πρόοδου του 2018 δίνει, έστα, δίνει έμφαση στην ανάγκη συλλογής περισσότερων δεδομένων για τα άσυλα, για τους ετούντες άσυλο, αλλά και για τη μετανάστευση. Είναι ανάγκη να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις αλλαγές στον τομέα αυτό της μετανάστευσης. Α, σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις της επιτροπές, α, σε σχέση με προηγούμενους κανονισμούς, προσφέρουμε αξιολόγηση και υπογραμμίζουμε το γεγονό ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα κενά στη στατιστική, στη συλλογή δεδομένων. Ποιοι είναι οι στόχοι μας. Βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να είμαστε πιο ακριβείς, πιο ενημερωμένοι και να έχουμε καλύτερη συχνότητα. Να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις επίουσες ανάγκες, να αυξήσουμε τη σταθερότητα των εθελοντικών στατιστικών στοιχείων και αυτοί να καταστούν υποχρεωτικοί ένας ε, στόχος επίσης είναι να μειώσουμε το, το βάρος ε, το οποίο αναγκάζονται να έχουν οι διάφορες εθνικές υπηρεσίες. Επίσης να αυξήσουμε την ευελιξία μας σε σχέση με μελλοντικέ ανάγκες. Η προτινόμενη τροπολογία του κανονισμού σε ό,τι αφορά καλύπτει αυτούς που ζητούν άσυλο για πρώτη φορά τους ανήλικους, τους μη συνοδευόμενους ανήλικους, περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις επανακαταστάσεις, καθώς και επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνθήκη στατιστικά στοιχεία για τη συνθήκη του Δουβλίνου, περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις επιστροφές και λεπτομερή στοιχεία για τις άδειες παραμονής. Οι ανάγκες αυτές στατιστικής βασίζονται σε διάφορες ε, συμβουλευτικές συζητήσεις που έχουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 2007 εισήχθησαν οι μέθοδος συλλογής δεδομένων και από τότε έχουμε συχνές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρατηρούμε τα όλα, και, είναι και αυξανόμενα κενά στη συλλογή δεδομένων. Είμαστε σε κοντινή επικοινωνία, σε στενή επικοινωνία με τις εθνικές αρχές, σε ιδιαίτερα στενή επικοινωνία με τους διευθυντές των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, καθώς επίσης και με την υπηρεσία έκδοσης ασύλου, αλλά και την Frontex, με διεθνείς οργανισμούς και με άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Α, αρκετοί εμπειρογνώμονες προσπαθούν να αναπτύξουν τον τομέα αυτών της στατιστικής την τελευταία δεκαετία και να μπορέσουν να καταστήσουν τα α, στατιστικά στοιχεία αυτά όλο και πιο σχετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανοίξω τώρα τη συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Ο Μπέγκετ Σίπελ έχει το λόγο. η οποία και δίνει το λόγο σε μια συνάδελφο που μιλάει εκ μέρους της, uh, της κυρίας Κιάνγκε. Τότε η Νάταλη Γκρίσπεκ θα έχει το λόγο, λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ε, Σοφή. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω ότι είναι ένα ε, κείμενο ευπρόσδεκτο, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και σε σχέση με την επικαιρότητα, αλλά και σε σχέση με την επιχειρησιακή οργάνωση των συστημάτων. Νομίζω ότι όπως μόλις μας εξηγήθηκε η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών είναι βασικό δεδομένο σε σχέση με ε, το, ε, το ζήτημα αυτό Ενδεχομένως αυτή η δουλειά των αξιωματούχων σύνδεσης μετανάστευσης ε, μπορεί να είναι μία ακόμη προσέγγιση που δεν είναι αρκετά ευρωπαϊκή, είναι πιο εθνική. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με την ίδια την οργάνωση, γιατί για την ώρα είναι πολύ συνδεδεμένη με, το, με τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ότι... Ε, με τη συνεργασία και με την Τζεσίλ και με τους υπόλοιπους συζητητέ. θα προσπαθήσουμε να προσδώσουμε έναν πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα ε, και στο κείμενο αλλά και στους στόχους που προσπαθεί να επιτύχει. Ούτω ή άλλω θα συζητήσουμε με του συναδέλφους όλο αυτό ε, το θέμα και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά ε, ώστε η δημιουργία αυτού του ευρωπαϊκού δικτύου να είναι αποτελεσματική ως προς τη μετανάστευση και θα ήθελα να πω επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό ε, σε σχέση με τη σύνδεση των διαφόρων υπηρεσιών. Ε, εχθές ήταν εδώ η κυρία Κατρίν Ντεμπόλ από την Ευρωπόλ. Το είπε και εκείνη κατά την ομιλία της ε, το σύνολο της οργάνωσης ε, ΕΑΖΟ, Frontex, ε, όλες οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο της λογικής αυτού του κειμένου ώστε να είναι αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα συνεργαστώ με τους εισηγητές και τους κοιόδης για το κείμενο αυτό. Η Κορνίλια Έρτς δεν είναι εδώ, οπότε η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Μετανάστευσης. Πρώτα να ακούσω τους εισηγητές, μετά ε, τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τεχνική απόψεω, ε, που εντάξει δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά η πράσινη είναι πλέον λίγο πιο πολυπληθή ομάδα από την ΚΟΕ. Οπότε κανονικά πρέπει πρώτα να μιλήσω εγώ. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να επικεντρωθώ στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και θα ήθελα να καταλάβω κάτι. Εχθέ ήταν εδώ ο Αυστριακό υπουργό Εσωτερικών ε, Εντάξει για, και μας μίλησε για ζητήματα ε, μετανάστευσης και έχω ε, κάπως μπερδευτεί. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει το επόμενο ήμιση του ε, έτους ή την περίοδο μέχρι τις ευρωεκλογέ για τα διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν κολλήσει και δεν προχωρούν. Συμφωνήσαμε για την επανεγκατάσταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις διαδικασίες και την οδηγία τη σχετική. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, πώς καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκβαση της Συνόδου πριν από δύο εβδομάδες που μίλησε για μια συνένεση εντός του Συμβουλίου για το Δουβλίνο. Ξέρουμε ότι αν το Συμβούλιο επιζητά συνένεση, ε, συνήθως ε, δεν, ε, δεν υπάρχει πουθενά το Κοινοβούλιο. Εχθές η Αυστριακή Προεδρία, όταν ερωτήθη σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες αποβίβασης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ε, εντάξει, τα συμπεράσματα λένε ότι πρέπει να κάνουμε έρευνα. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν σας ζητώ να ολοκληρώσετε γρήγορα αυτή την έρευνα, αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα, να μας δώσετε μια καλύτερη εικόνα, εκτός από τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε, πού πηγαίνουμε με, τη γενικό, με το γενικότερο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Έλστρα δεν είναι εδώ. Η Σίδρια, η κυρία Κιέγκε δεν είναι εδώ. Και η κυρία Κινίτσου θα διαβάσει μια δήλωση εκ μέρους της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θα πάρω το λόγο από πλευράς της κυρίας Κιέγκε, η οποία είναι σε μία αποστολή παρατήρηση εκλογών. Καταρχάς, ε, ζητώ συγγνώμη ε, από όλους για την ε, εκ της, για την απουσία της. Ευχαριστεί λοιπόν η κυρία Κέγκε την Επιτροπή για την παρουσίαση και για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για τους ε, συνδέσμους. Ήδη το 2015, όταν συζητήσαμε την, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, η Κομισιόν είχε ήδη τονίσει ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστό μείγμα μεταξύ πολιτικής στο εσωτερικό της Ένωσης και στο εξωτερικό. Και τότε όλα τα κράτη-μέλη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι τρίτες χώρες κλήθησαν να εργαστούν όσο καλύτερα μπορούν για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν καθοριστεί με τα κράτη-μέλη και για να υπάρξει η βέλτιστη διαχείριση στα πλαίσια της μέγιστης προστασίας ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθερών. Οι σύνδεσμοι αυτοί για τη μετανάστευση ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. Όπως όμως και η Κομισιόν τονίζει στην πρότασή της, ε, ε, οι δυνατότητες που μας παρέχουν δεν ε, υλοποιήθησαν πλήρως. Υπάρχουν προβλήματα στην ανταλλαγή προφοριών, στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και γενικότερα στη διάδοση της ενημέρωσης. Η κυρία Κέγκε θεωρεί ότι 500 τέτοιοι σύνδεσμοι που έχουν αποσπαστεί σε τρίτες χώρες και το δίκτυό τους αποτελεί μια δυνατότητα που εάν βελτιωθεί ε, μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη διαχείριση της μετανάστευσης. Σημερίζεται τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απλώς θα υποβάλει κάποιες τροποποιήσεις για να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταλλαγή προφοριών και ούτω ώστε να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα ιδιαίτερα των πλέον ευαλώτων ατόμων και να εφαρμόζεται η αρχή ε, των μη διακρίσεων και της μη επανεισδοχής. Σας, ε, της μη επαναπρόθεσης καλύτερα. Ευχαριστώ. Αυτά από πλευρά τη κυρία και η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ. Στρέφομαι στην Επιτροπή και την ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνατε σήμερα το πρωί και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη ε, που επέδειξαν προς εμένα ως εισηγήτρια για το θέμα των στατιστικών για τη μετανάστευση. Προσβλέπω όπως πάντα στη στενή συνεργασία με όλους και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι στατιστικές για τη μετανάστευση δεν είναι τόσο ε, ελκυστικό θέμα όπως για παράδειγμα ο κανονισμός του Δουβλίνου ή οποιοδήποτε άλλο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο παραποτέ να έχουμε πιο στοιχειοθετημένη αντιμετώπιση του θέματος ε, ασύλου και μετανάστευση. Και για να έχουμε λοιπόν ε, τα απαραίτητα στοιχεία χρειαζόμαστε και τις κατάλληλες στατιστικές που ανακαλύπτουν όλους τους τομείς. Κατά τη γνώμη μου, η πολιτική, και ελπίζω να συμφωνούμε όλοι, η πολιτική θα έπρεπε στο μέτρο του δυνατού να βασίζεται σε στοιχεία και επιστημονικές αποδείξεις. Άρα πρέπει να είμαστε, πιστεύω, ιδιαίτερα ρεαλιστές. Αντιμετωπίζοντα το θέμα αυτό και ανεξάρτητα από τις απόψει που μπορεί να υπάρχουν στην Ευρώπη για την μεταναστευτική πολιτική όλοι, πραγματικά όλοι, θα έπρεπε να έχουμε ένα στόχο. Να έχουμε πραγματικά αξιόπιστες στατιστικές για να καταλάβουμε τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή εξετάζω την πρόταση της Επιτροπής και μαζί με τους κοιόδης θα τη μελετήσουμε αναλυτικά Ήδη σήμερα. Δεν θα προκαταλάβω σήμερα το σχέδιο έκθεσης, αλλά από την έρευνα που έχουμε κάνει για το θέμα φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη συλλέγουν πολύ περισσότερες στατιστικές από αυτές που αποστέλουν στην ε, Eurostat. Και πολλοί, ε, ναι μεν, στέλνουν ε, σε μη τα στατιστικά του στοιχεία και τα δημοσιεύουν σε εθνικές εκθέσεις. Άρα, Πολλά από τα στοιχεία αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Νομίζω ότι χρειάζεται επίσης ε, να έχουμε πληροφορίες σε πολύ πιο αναλυτικό επίπεδο με βάση και συμπληρωματικά κριτήρια για να έχουμε επαληθεύσιμες στατιστικές χωρίς να αυξηθεί η γραφειοκρατία για τα κράτη-μέλη. Η πρόθεσή μου είναι να σας υποβάλω ένα σχέδιο έκθεσης ε, πριν τις 10 Σεπτεμβρίου για να το συζητήσουμε στη συνεδρίασή μας στις 27 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία για τις τροπολογίες θα είναι 4 Οκτωβρίου και στοχεύω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ως Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου και για να λάβουμε κατά την μήνυ ολομέλεια τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου διαπραγματευτική εντολή για τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι είναι αρκετά σφιχτό το χρονοδιάγραμμα αλλά θα μας αφήσει κάποιε δυνατότητε τριμερού διαλόγου κατά τη διάρκεια τη τρέχουσα θυσία. Αυτό βεβαίω, εφόσον το Συμβούλιο πραγματικά θέλει να προωθήσει το θέμα αυτό και να συζητήσει μαζί μα. Είμαι πεπισμένη ότι εμεί από την πλευρά μα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εξέτασή του. Σα ευχαριστώ πολύ. Ωραία, λέει πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε λίγο καθυστερήσει. Ε, άλλα τέσσερα άτομα έχουν στήσει το λόγο. Σταχόφσκι, Βεργιά, Μιράντα και Λόπεθ Αγγιλάρ. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ ο καθένας και μετά θα επανέλθω πολύ σύντομα προς την Επιτροπή για να μας απαντήσει ερωτήσεις που θα μπορούσαν να έχουν. Και μετά θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σταχόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συζητητές και την Κομισιόν. Θα σας παρουσιάσω την άποψη κυρίας Μουσολίνη. Η οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες επιτέλους ε, διατύπωσαν την άποψη ότι χρειάζεται συνδυασμός της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης με βάση προβλέψιμη και λογική διατύπωση κανόνων και σε μια διαθρωμένη συνεργασία και συντονισμό με τις χώρες ε, προέλευσης και ε, μετάβασης. Οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να συμμετέχουν ε, σε έναν επικοδομητικό διάλογο με τις τρίτες χώρες. Αυτό είναι προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και η διακίνηση. Για τις στατιστικές τονίζω αυτή είναι η δική μου άποψη ότι χρειαζόμαστε αξιόπιστα στατιστικέ. Και μία ερώτηση προ την Επιτροπή. Τι γίνεται στη Σουηδία. Αναφέρεται η έκθεσή σα στα γεγονότα στο Μάλμε. Αυτέ οι συμμορίε και διάφορα άλλα. Πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βεργιά. Σας ευχαριστώ που επιτρέψατε στους ε, διερμηνείς να διαβάσουν το μήνυμά τους και τους σέβεστε, γιατί δεν γίνεται συχνά. Είμαι η συγγήτρια για τα δύο αυτά κείμενα και όπως και η Κονέλια Ένς δεν είναι, θα έπρεπε να μιλήσω εκ μέρους της ε, συντονίστρια. Ξέρω ότι έτσι καταναλώνω το χρόνο ομιλίας, αλλά επί της μεθόδου, σε μία ώρα να θέλουμε να συζητήσουμε για δύο νέε νομοθετικές προτάσεις και για την έκθεση πρόοδου για τη μετανάστευση δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος εργασίας αλλά ε, όλο και πιο σύνηθε εδώ. Λοιπόν, τάχιστα. Το θεματολόγιο μετανάστευσης. Θέλω να επανέλθουμε στο 2015 όταν εγκρίθηκε αυτό το θεματολόγιο είχε τέσσερις άξονες σε σχετική ισορροπία μεταξύ τους. Και σήμερα τι έχει γίνει. Αν δούμε τον απολογισμό σήμερα, ασχολείται μόνο με την λεγόμενη παράτυπη μετανάστευση. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τι προσέγγιση είναι αυτή. Και εμείς εδώ μέσα ως κοινοβούλιο. Γιατί ε, αποκλειστικά ασχολούμεθα με αυτή τη διάσταση. Ενώ λέμε ότι θέλουμε ολιστική προσέγγιση. Ενώ θέλουμε να υπάρξει και εσωτερική και εξωτερική αντιμετώπιση. Οι διαδρομές που αναφέρονται είναι μόνο οι παράτο, παράτυπες διαδρομές. Δεν είναι σωστή αυτή η μέθοδος ε, αντιμετώπισης του θέματος. Και καταγγέλλω για άλλη μια φορά, γιατί δεν έχει γίνει από κανέναν, για άλλη μια φορά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης για το καταπίστευμα για την Αφρική. Ωραίε και στατιστικές. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με την κυρία Βίξτρεμ, γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλές στατιστικές και αν έχουμε καλές στατιστικές θα καταφέρουμε να διαψεύσουμε μια σειρά από ψεύδι που λέγονται. Η Γκουε δεν είχε αρκετό χρόνο. Πρόεδρο, μα τόσο χρόνο έχουμε. Δεν ξέρω, αν θέλετε μπορούμε να κάτσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά αυτό ο χρόνο είχε προβλεφθεί. Παρακαλώ τους άλλους συναδέλφους που μπαίνουν να σεβαστούν λιγάκι τους ομιλητές για να τελειώνουμε και να ψηφίσουμε. Η κυρία Μιράντα, 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω για κάτι που έγινε την ε, περασμένη εβδομάδα. Τις στατιστικές για τους νεκρούς. Μετράνε νεκροί. Τα άτομα που δεν διασώζονται. Ε, τα έχετε καθόλου στο μυαλό σας ε, κύριοι και κύριοι στις Επιτροπές. Αυτός ο συντονισμός των ε, μεταναστευτικών πολιτικών θα ασχοληθεί με τα κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, όπως η Μάλτα που δεν θέλουν να ε, αποβιβαστούν ε, τα διασωθέντα άτομα στα λιμάνια τους την προηγούμενη εβδομάδα. Το σκάφος Open Arms με ισπανική σημαία δεν μπόρεσε να ελιμενιστεί στα λιμάνια της Ιταλίας και της Μάλτας. Εμείς ήμασταν εκεί μέσα σε αυτό το σκάφος και το διαπιστώσαμε. Καλά τα λόγια και οι παρουσιάσεις και η νομοθεσία άριστα. Αλλά οι στατιστικές για τους νεκρούς δεν αναφέρονται πουθενά. Και θα ήθελα μια απάντηση από πλευρά της Κομισιόν. Γιατί επικοινωνήσαμε, επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε κατά τη διάρκεια του διάπλου και δεν μας απάντησε κανείς. Πώς είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται σε ευρωπαϊκά σκάφη να πιάσουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Αυτό είναι ντροπή. Και έτσι ξεφτυλιζόμαστε όλοι. Και εμεί οι βουλευτέ και οι θεσμοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή. Τη συζητάμε, το συζητάμε αυτό το θεματολόγιο για τη μετανάστευση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και ιδιαίτερα στην τελευταία ολομέλεια το συζητήσαμε. Άρα σχολιάστε παρακαλώ τα τέσσερα σημεία που αναφέρθηκαν στις συζητήσεις που κάναμε στην προηγούμενη ολομέλεια στο Στρασβούργο. Τα οποία είναι πρώτον αποβιβάσεις, λιμένες αποβίβασεις. Εφόσον σέβονται το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, Πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσουν αν δεν έχουμε διμερεί συμφωνίες για να μπορεί να συμβεί αυτό με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Οδηγείται η διευκόλυνση. Ζητήσαμε την τροποποίησή της, ούτω ώστε να μην ποινικοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια και η διάσωση στις ανοιχτές θάλασσες. Τρίτον, η πλειοψηφία του σώματός μας ζητάει νόμιμες ε, Δυνατότητε μετανάστευση. Αν δεν υπάρχουν νόμες δυνατότητε, τότε μιλάμε μόνο για παράτυπη μετανάστευση. Γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα νόμιμη μετανάστευση. Και τέταρτον, η εθελούσια αλληλεγγύη δεν είναι αλληλεγγύη. Και δεν έχει να κάνει με την εντολή που αναφέρεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να υπάρξει δεσμευτική αλληλεγγύη για όλα τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο για του ε, επιθυμούντε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να επανέλθουμε στην Επιτροπή. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα η έκθεση πρόοδου που είναι μια ενιαία έκθεση ήδη από την εισαγωγή λέει ότι παρουσιάζει μια γενική εικόνα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ολόκληρο το θεματολόγιο. Γι' αυτό και είναι μια κοινή έκθεση και δείχνει κατά πόσο θα πρέπει να είναι καθολική η δουλειά που κάνουμε. Χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία. Την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ό,τι αφορά την μετανάστευση αλλά και την ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας είναι ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Επίσης το ίδιο λέμε και εκεί που περιγράφουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε προστασία των εξωτερικών συνόρων, εσωτερική συνεργασία εξακολουθούμε να παρακολουθούμε όλα αυτά τα ζητήματα αξιών, βασικών αξιών. Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις για το άσυλο, αλλά και την αξιολόγηση υπαρχιακής, ε, περιφερειακής με συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, σε ό,τι αφορά το άσυλο στην παράγραφο 12 υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σε σχέση με την παρούσα κατάσταση αλλά και τα μελλοντικά βήματα. Είναι ανάγκη να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος ώστε να περιοριστούν τα θέματα προς διαπραγμάτευσης και νομοθετικά ζητήματα πιο συγκεκριμένα που περιλαμβάνονται και στον κανονισμό του Δοβλίνου και περαιτέρω ζητήματα που αφορούν την χορήγηση ασύλου. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας από κοινού μαζί με το Συμβούλιο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συμπεράσματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Θα έχουμε μια έκθεση πρόοδου και τον Οκτώβριο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει η Πρόεδρος, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει η κυρία Ντολφίνο. Δεν υπήρχαν ερωτήσεις. Ο κύριος Βρόνσκι ίσως. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ευχαριστήσω για την υποστήριξη του συναδελφού. Δεν πιστεύω ότι απαντήθηκαν οι ερωτήσεις. Θα επιστρέψουμε όμως αυτά τα ζητήματα ούτως ή άλλως, γιατί αυτή είναι απλά η έναρξη της διαδικασίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία τώρα, Πρωτού έρθει ο Επίτροπος Κίνγκ. πρώτη ψήφος ό,τι αφορά την ομιμοποίηση του χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων από τη χρήση τους από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Επίσης εγκρίνεται. κυρία Γκρίσπετ, αμοιβαία αναγνώριση δέσμευσης και δίμευσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε. Επίσης εγκρίνεται με ευρία, πλειοψηφία. Και τέλος, το προσέδιο για τη Eurojust. Άρχεται η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Okay, so we've we've made up <laughs> we've made up for lost. Καταφέραμε να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, τον ανοιχτό διάλογο της ΛΥΜΠΕ με τον Επίτροπο Κίνγκ. Να ζητήσω από τους συναδέλφους να επιστρέψουν στη θέση τους. Ο Επίτροπος είναι εδώ και θα ξεκινήσει την ομιλία του. Να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο King για, την, για τον τρίτο ανοιχτό διάλογο σε θέματα ασφαλείας και εφαρμογή της αποφασής των αποφάσεων Προύμ και το αγαπημένο μου ζήτημα PNR, καταγραφή επιβατών. Μια ταχεία εισαγωγή. Έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Στις 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μια προπαρασκευαστική συνάντηση όπου η έκθεση του καθηγητή του παρουσιάστηκε. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφα της έκθεσης αυτής με τη συμμετοχή όχι μόνο της Επιτροπής αλλά και του Συμβουλίου καθώς και εμπειρογνώμων από τη Γερμανία και την Ισπανία αλλά και η μελέτη του καθηγητή του επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών υπογραμμίζοντας την δυσκολία αξιολόγηση των δεδομένων αυτών λόγω των στατιστικών στοιχείων που λείπουν και δεν επιτρέπουν την ορθή ανταλλαγή με σκοπό βεβαίω την πρόληψη του εγκλήματος. Κάτι το οποίο δυσκολεύει την αξιολόγηση της επιμέρους αξίας που προσθέτει η ανταλλαγή δεδομένων. Η γραμματεία του Συμβουλίου η προθεσμία ήταν 28 Αυγούστου του 2011 7 χρόνια πριν. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι απολύτως λειτουργικά με διαφρονιδών δεδομένα. Η γερμανική BKA υπογράμμισε την σημασία και την ανάγκη των, της ανταλλαγής δεδομένων και είπε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, αλλά λόγω έλλειψης πόρων ε, δυσκολεύεται η εφαρμογή τα βήματα που πρέπει να κάνουμε καλούν για περαιτέρω νομική βοήθεια. Η Επιτροπή σε σχέση με την εφαρμογή του PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 κράτη-μέλη έχουν δηλώσει ότι χρησιμοποιούν την οδηγία αυτή. Η Επιτροπή έχει λάβει 20 ειδοποιήσεις από κράτη-μέλη σύμφωνα με τις οποίες θα εφαρμόσουν την οδηγία για τις εσωτερικές πτήσεις. αρκετά κράτη-μέλη έχουν ε, διάφορες απορίες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προυν. Δύο κράτη-μέλη. Ελάχιστα. αρκετά μέλη αμφισβήτησαν κατά πόσο η οδηγία PNR είναι συμβατή με το δικαστήριο αλλά και τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορούν τις πτήσεις ε, τα ιδιωτικά αεροπλάνα. Επίτροπε, έχετε 15 με 20 λεπτά πάνω στο ζήτημα των δεδομένων ΠΡΟΥΜ και PNR. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ, χαίρομαι που σας βλέπω. Πάντα χαίρομαι. Πάντα χαίρομαι που είμαι δίπλα σας και χαίρομαι που έχω δυνατότητα να σε ενημερώσω για κάποια στοιχεία που αναφέρατε, για τα τελευταία, τελευταία εκδοχή τους δηλαδή. Όπως είπα, πάντα χαίρομαι για τη δυνατότητα συνέχισης του διαλόγου για τις προσπάθειες που κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια ένωση ασφαλείας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε για οποιαδήποτε πλευρά του θέματο αυτού, είτε τώρα είτε όταν θα μιλήσουμε το Σεπτέμβριο, στι αρχέ Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια του διαθρομένου διαλόγου για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, να αντιμετωπίσουμε τι μεθόδου που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτε, όπλα, ε, εκρηκτικά, η χρηματοδότησή του. και προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μα για να βελτιώσουμε την προστασία των δημοσίων χώρων, να αντιμετωπίσουμε την ρίζοσπαστικοποίηση στις κοινότητες μας, στις κοινωνίες μας, στις τοπικές κοινωνίες και στο ίντερνετ η ενίσχυση της, ε, πολιτικής, της αστυνομικής συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, η αντιμετώπιση των κύβερνων απειλών για να εφαρμοστεί η οδηγία νης για να ολοκληρωθεί η εργασία γύρω από την κυβερνοασφάλεια, η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, ζωτικό θέμα για την ευρύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων προστασίας ή για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκλογών. Όλα αυτά τα θέματα με χαρά να τα συζητήσω. Ζητήσατε όμως να εστιάσω στην εφαρμογή και κατάσταση πραγμάτων για την οδηγία για το PNR και τις αποφάσεις του ΠΡΙΜ. Με χαρά να αναφερθώ και σε αυτά. Θεμελιώδη θέματα είναι αυτά τη δουλειά μα για να ενισχύσουμε την ανταπόκριση τη Ένωση στην τρομοκρατία, το σοβαρό έγκλημα και τις κύβερνο απειλές. Βασικό στοιχείο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και τα στοιχεία για την εφαρμογή που σας απασχολούν ιδιαίτερα όπως και εμένα. παραλαμβάνω. για να υπάρξει ουσιαστικό πλαίσιο της Ένωσης Ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και πρέπει να αξιοποιούμε πλήρως τα ήδη υπάρχοντα μέσα και τις, ε, να εφαρμόζουμε τις ληφθήσεις αποφάσεις. Όπου δεν γίνεται αρκετά αυτό πρέπει να γίνεται. Η οδηγία για το PNR είναι συστατικό στοιχείο της προσπάθειάς μας. Η επεξεργασία των στοιχείων PNR θα ενισχύσει την ε, ανταπόκρισή μας στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Κανένα άλλο εργαλείο δεν μας επιτρέπει να εντοπίσουμε αγνώστους υπόπτους όπως η ανάλυση των στοιχείων του PNR. Για παράδειγμα βλέπουμε που γίνονται ύποπτα ταξίδια Και έτσι αντιμετωπίζουμε το σοβαρό έγκλημα και την ενεργό τρομοκρατία. Όπω ξέρετε, αυτή η οδηγία εγκρίθηκε σε ενωσιακό επίπεδο μετά από μακρόχρονη και ιδιαίτερα ε, επίμαχη διαδικασία. Άρα πρέπει τώρα που εγκρίθηκε οπωσδήποτε να το αξιοποιήσουμε. Να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το ισχυρό μέσο. Όπως μόλις ακούσατε, προθεσμία για τα κράτη-μέλη ή προθεσμία για να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη αυτή την οδηγία ήταν 25 Μαΐου. Μέχρι τώρα, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, τα 15 κράτη-μέλη έχουν ενημερώσει επισήμω την Κομισιόν για τα μέτρα που έχουν πάρει για να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία. Το γεγονό ότι δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη με ανησυχεί. Αλλά πιστεύω ότι και άλλα κράτη-μέλη θα ολοκληρώσουν τις επόμενες εβδομάδες τη διαδικασία. Και φυσικά ε, τους παρακολουθούμε. Κάποια κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει λιγότερο τη διαδικασία εφαρμογή από άλλα, αλλά όλα τα κράτη-μέλη, κατά τη γνώμη μου, δεσμεύονται στη μεταφορά της οδηγίας αυτής και προσπαθούν να αναπτύξουν τα εθνικά συστήματα PNR, η πληροφόρηση που έχουμε από τα κράτη-μέλη, καταδεικνύει ότι ήδη έχουμε από τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Για παράδειγμα, τον περασμένο Απρίλιο πήγα στην Βελγική υπηρεσία μόνο τρει μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματός τους και είχαν συγκεκριμένε επιτυχίε για περιπτώσεις ε, μεταφοράς ε, μετρητών, ε, διακίνηση ναρκωτικών και ξένων μαχητών. Άρα τα κράτη-μέλη που βραδιπορούν ε, στερούνται ενός τόσο σημαντικού μέσου. Και μειώνεται όμως και ο ενωσιακός μηχανισμός PNR συνολικά. Δυσχεραίνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά από το Europol με βάση τις συνθήκες που καθορίζει η οδηγία. Ο μηχανισμός αυτός είναι όσο ισχυρός είναι ο πιο αδύνατος κρίκος του. Επίσης, μειώνεται μέσω της εφαρμογής της, μάλλον λόγω της καθυστέρησης εφαρμογής της, μειώνεται και η νομική ασφάλεια για τις εταιρείε, τις αεροπορικές εταιρείε και είναι επιζήμια και ε, για τους ταξιδιώτες, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν ε, την ίδια προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη τα τελευταία δύο χρόνια. Πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν. Τους δώσαμε και χρηματοδότηση και εμπειρογνώμονες, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών σε πολλές περιπτώσεις. Ανταλλάξαμε σημειώματα πριν ε, την συνάντηση αυτή, όπου αναλυτικά αναφέρουμε τα μέτρα στήριξης προς τα κράτη-μέλη που έχουμε δώσει. Επίσης ε, προτείνουμε και ενθαρρύνουμε και την ανταλλαγή στοιχείων μέσω ομοτήμων, ούτως ώστε αυτοί που έχουν περισσότερη ε, εμπειρία να βοηθούν τους βραδιπορούντες. Και θα συνεχίσουμε να προτείνουμε όλες αυτές τις μεθόδους βοηθείας. Παράλληλα, θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή. Αυτό είναι το καθήκον μας και ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μέσω, εάν χρειαστεί, εκκίνησης διαδικασιών επί παραβάση. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την εφαρμογή, ούτω ώστε ήδη αυτό το μήνα να αναλυφθεί δράση κατά των κρατών μελών που μέχρι τούδε δεν μας έχουν ενημερώσει για το τι έχουν κάνει για τη μεταφορά αυτής της οδηγίας που είναι τμήμα και της ευρύτερη προσπάθειάς μας για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εφαρμογής του νόμου. Υπάρχουν δύο πιλωτικά προγράμματα που κάναμε ήδη για να δούμε πώς όλες αυτές οι υπηρεσίες στα κράτη-μέλη μπορούν να ανταλλάξουν αυτά τα στοιχεία. Και η Europol συμμετέχει πλήρως σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα έχουμε 16 τέτοιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο της Europol και μπορούν να ενημερωθούν για αυτά τα στοιχεία. Επίση, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να έχουμε ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών για την εφαρμογή τη οδηγία. Με στόχο και πάλι τη μέγιστοποίηση του ωφέλου. Τώρα για το πριμ. Η ανταλλαγή προφοριών πιστεύουμε και εσεί πιστεύετε ότι είναι βασικό στοιχείο τη συνεργασία των αρχών εφαρμογή του νόμου στα πλαίσια τη Ένωση Ασφαλεία. Και αποφάσει του πριμ παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Όπω σωστά είπατε, στα πλαίσια τη τελευταία δεκαετία που υπάρχουν αυτέ οι αποφάσει, το ΠΡΙΜ απέδειξε ότι είναι χρήσιμο εργαλείο για τη συνεργασία αυτών των αρχών. Βοήθησε να διαλευκανθούν εγκλήματα. Η χρήση του από χρόνο σε χρόνο αυξάνεται και η ενημέρωση που μα δίνουν τα κράτη-μέλη είναι ότι εκτιμούν ιδιαίτερα αυτέ τι δυνατότητε. Σα δώσαμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του πριμ λοιπόν ήδη. Αλλά οι αποφάσεις του πριμ δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη. Παρά το ότι η Κομισιόν έδωσε και τεχνική οικονομική βοήθεια και διευκόλυνε την ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών. Μεταξύ του 2008 και του 2013 η Επιτροπή έστειλε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με το ΠΡΙΜ. Και στα πλαίσια του Ταμείου Εσωτερική Ασφαλεία προβλέπονται 22 εκατομμύρια προς αυτή την κατεύθυνση και άλλα 3 εκατομμύρια για να στηρίξουμε την εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών ε, στοιχείων συλλογής, ε, συλλογής στοιχείων από εγκλήματα. Επίσης, κάποια κράτη-μέλη δεν φύρμωσαν εγκαίρως τη διαδικασία και οι διαδικασίες παραβάσει υπάρχουν κατά κρατών μελών, αλλά και τα τέσσερα αυτά κράτη έχουν σημειώσει πρόοδο. Άρα καλό είναι να συζητήσουμε τώρα για το μέλλον του πριν. Τι μορφή θα μπορούσε να έχει. Οι αδυναμίες έχουν να κάνουν με μακροχρόνιες διαδικασίες για ε, πληροφορία για το τι γίνεται όταν εντοπιστεί κάποιος. Και έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια και στην ιατροδικαστική και στην τεχνολογία γενικότερα πρόοδους που θα πρέπει να παίξουν ρόλο στο πώς θα προσαρμόσουμε το πριν. Και επίσης έχει αλλάξει φυσικά και το καθεστώ για την προστασία δεδομένων. Όπω λέει και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η Κομισιόν μέχρι τον ερχόμενο Μάιο θα εξετάσει τι αποφάσει πριν για να τι ευθυγραμμίσει με αυτή την οδηγία. Και αν χρειαστεί θα κάνουμε τι προτάσει για την τροποποίηση αυτών των αποφάσεων. Θα εξετάσουμε και την αναγκαιότητα, αναλογικότητα και τεχνική δυνατότητα νέων τεχνικών λύσεων. Η Επιτροπή θα κάνει μια μελέτη αντικτύπου συγγνώμη, μια μελέτη εφικτότητα που θα ξεκινήσει του επόμενου μήνες σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και άλλους εμπλεκομένους. Και θέλω να πω επίσης ότι τα αποτελέσματα από την έκθεση που έχουμε για την ανταλλαγή στοιχείων DNA είναι σημαντική συμβολή σε αυτή την εργασία. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι γνωστά αρχές του επόμενου χρόνου. Τώρα, κάτι ακόμη για τους άλλους δύο πυλώνες της εργασίας μας για περισσότερη και ευφιέστερη ανταλλαγή στοιχείων για την ασφάλεια και διαχείριση των συνόρων. Πρώτα απ' όλα να καλύψουμε τα κενά στην ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και ιδιαίτερα την κυρία Γκάλ που ήταν η συγκήτρια και τους κοιόδης ε, για την υπερψήφιση του συστήματος αιτιάς την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια μαζί με τη συμφωνία για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Πιστεύω ότι τα συστήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ούτω ώστε οι πολίτε μα να είναι ασφαλεί, όπω και τα σύνορά μα. Επίση, ψηφίσατε την ενίσχυση του οργανισμού Ιγιου e λίσα Ευχαριστώ την εισηγήτρια κυρία Μακοβέη και τους Κιώδη. Έτσι θα συνεχίσουμε να εξυγχρονίζουμε τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών εφαρμογής του νόμου και διαχείριση των συνόρων. Το EU Λίσα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δεύτερον, διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων συλλογής πληροφοριών που έχουμε. Το έχουμε ήδη συζητήσει, θα το συζητήσουμε και περαιτέρω σε λεπτομέρεια, πιστεύω. Η Επιτροπή σα τον Ιούνιο ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και θίξατε μια σειρά από θέματα. Δεν υπήρχε χρόνο τότε να απαντήσω, τουλάχιστον πλήρω. Έστειλα μια επιστολή στον ε, πρόεδρο Κλόντ Μωράες και ελπίζω η επιστολή μου να ε, ικανοποίησε κάποια, κάποιες ερωτήσεις που είχατε θέξει και εσείς συγκεκριμένα κυρία Πρόεδρε. Αλλά εάν δεν έχει απαντηθεί, δεν έχουν απαντηθεί όλα, ευχαρίστω να απαντήσω και σήμερα. Βέβαια, η προστασία των ε, πολιτών μας πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως ξέρετε, υπάρχει και ο αντίστοιχος φορέας και ο επόπτης προστασίας δεδομένων στις νέες μας προτάσεις. Και καταλαβαίνω βεβαίως την επιθυμία και των εισηγητών και της Επιτροπής να υπάρξει ταχεία πρόοδος, στη, να υπάρξει ταχαίως η εξέταση αυτών των, των προτάσεων. Ελπίζω οι τριμερείς συζητήσεις να αρχίσουν ε, σύντομα μετά τις διακοπές. Και ελπίζουμε αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει μέχρι τέλο του χρόνου. Και επίση, η βελτίωση τη ανταλλαγή πληροφοριών είναι στοιχείο κλειδί στην προσπάθειά μα για μια αποτελεσματική ένωση ασφαλεία. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία μα τα τελευταία χρόνια. Έχει πιστεύω συμμεθεί πρόοδο, αλλά πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν και πρέπει να τα κάνουμε ε, συμβαδίζοντας πλήρως και συνεργαζόμενοι στενά με σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα οι συντονιστές. Η κυρία Μέτσολα βέβαια δεν είναι εδώ, οπότε η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Έχω μια σειρά από ερωτήσει. Πολύ συχνά για θέματα ασφαλείας μας λέτε δεν κάνουμε αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Αλλά αν κοιτάξω τα στατιστικά στοιχεία ποινικών αδικημάτων διαπιστώνονται σε πολλούς τομείς είτε είναι στάσιμα, είτε είναι στάσιμα τα αδικήματα αυτά, είτε σε άλλους τομείς μειώνονται. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Γιατί λέμε ότι δεν κάνουμε αρκετά. Πολλά έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά εφαρμόζονται μερικά ή καθόλου. Πώς μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν ότι δεν επαρκούν τα μέτρα που έχουμε ήδη εγκρίνει. Αναφέρατε το PNR ότι έτσι ε, εντοπίζουμε αγνώστους ε, υπόπτους. Χρειάζονται ε, και πολύ πόροι και πολύ προσωπικό για να τα συλλέξουμε όλα αυτά που δεν έχουμε αλλού. Αλλά, όπως ξέρετε, η αρχική αιτία για την οποία αναπτύξαμε αυτό το σύστημα ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε κάνει τίποτα. Είπατε ότι σε μία περίπτωση στο Βέλγιο είχαμε καλά αποτελέσματα. Είπατε ότι για ναρκωτικά και για τρομοκρατία είχατε αποτελέσματα. Τι εννοείτε, συνελήφθη κανεί ή απλώς παρακολουθούμε κάποιους υπόπτους. Πιο συγκεκριμένα παρακαλώ. Τώρα για το πρωίμ. Με καταπλήσει. Όταν ακούω πόσα εκατομμύρια, πόσα χρόνια έχει πληρώσει μόνο η Ένωση. Και ε, ακόμη δεν λειτουργεί. Και πέρα από όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχει δαπανίσει μέσω της Κομισιόν ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος, υποθέτω ότι και τα κράτη-μέλη έχουν και εκείνα δαπανίσει περισσότερα. Πώς αξιοποιούμε την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτήσεών μας. Ω φορολογούμενο, αν ακούω ότι μόνο η Ένωση έχει δώσει 50 εκατομμύρια και ακόμη δεν λειτουργεί, τότε αυτό είναι κατασπατάληση του χρήματο των φορολογουμένων. Τώρα για την παραπληροφόρηση. Μα τι είναι πλέον παραπληροφόρηση να ρωτήσω, τι είναι ψεύτικες ειδήσει. Έχετε κάποιο αφιορισμό, έχετε κάποια αντίληψη για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι είναι ψεύτικες ειδήσει και πόσα στοιχεία χρειάζεται να συλλέξουμε για να το αποφασίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Λείπει η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Κίνγκ που είναι μία ακόμη φορά μαζί μας για να μας παρουσιάσει την ενημέρωση αλλά και να απαντήσει και στα ερωτήματά μας. Ευχαριστούμε και για το χιούμορ σας σε σχέση με την, ε, ε, το μακροχρόνιο της διαδικασίας για να καταλήξουμε σε ένα PNR. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μας ήθελε ένα PNR ευρωπαϊκό, ένα και μοναδικό εργαλείο, όχι 27-28 PNR. Τουλάχιστον για τη δική μου ομάδα ε, θα επιθυμούσαμε και μια υποχρεωτική υποβολή δεδομένων ήταν πάρα πολύ βέβαια η ενδιαφέρουσα και επικοδομητική ε, η παρουσίασή σας. Είπατε ότι ήταν και πάρα πολύ επίγον. Θα θυμάστε ότι είχαμε μπλοκάρει όλο το σύστημα και κάποια χρόνια μετά έχουμε 15 κρατημέλη που έχουν PNR. Ένα σύστημα το οποίο βέβαια προσφέρει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά ε, ζητήματα προστασίας και ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες παραμένει ωστόσο ένας μηχανισμός ε, ατελής κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι τόσο ευρωπαϊκός ε, όσο θα ήθελε η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και που μας εξηγήσατε σήμερα το πρωί. Το ζήτημα των τσάρτερ όμως ε, με απασχολεί εμένα. Η έλλειψη δεδομένων ε, όσων οργανώνουν, για παράδειγμα, εγκληματικές δραστηριότητες ή τρομοκρατικές επιθέσεις και μπορούν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω των τσάρτερ, να παρεκκλίνουν, ε, να παρακάμψουν το PNR. Ε, θα περίμενε κανείς τα μεγάλα αεροδρόμια να προστατεύουν ε, τα δικαιώματα των, ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Τα μικρά όμως αεροδρόμια ε, αποτελούν ένα κενό στο σύστημα. Ε, μία ακόμη ερώτηση τώρα για να ολοκληρώσω. Όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας που αφορούν την υποβολή, την εθελοντική δεδομένων, όσον αφορά τα Τη πτήση μεταξύ των κρατών μελών. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, πώς εξελίσσεται και πώς λαμβάνεται υπόψη αυτό από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που μακρηγόρησε. Κυρία Σαρτζεντίνη, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τη διαφορά ε, του PNR ε, ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά και του δικού μα PNR, αυτό το ζήτημα Ευρωπαίοι πολίτες φτάνουν στον Καναδά και μετά φεύγουν από εκεί, αναχωρούν από εκεί. Αν δεν υπάρχει κάποιος εντοπισμός κινδύνου, τότε πρέπει τα στοιχεία τους από τη βάση δεδομένων να διαγράφονται. Αυτό ζητούμε. Παρά, παρόλα αυτά, αυτή είναι τουλάχιστον ε, η άποψη του Ιουλίου του 2017 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρόλα αυτά, το δικό μα PNR δεν το προβλέπει αυτό. Πώ είναι δυνατόν να ε, ξεπεράσουμε αυτέ τι δύο δυσκολίε. Πραγματικά είναι τρομερά υποκριτικό αυτό. Ζητούμε από τον Καναδά να διαγράψει τα δεδομένα από τη δική του βάση δεδομένα, αλλά εμεί δεν το κάνουμε αυτό. Πώ θα το υπερβούμε αυτό, αυτήν την άδικη κατάσταση. Και όσον αφορά τώρα την απόφαση του Συμβουλίου για το ε, ΠΡΟΥΜ. Είναι μια απόφαση του 2018, είναι, πα, είναι πεπαλαιωμένο το κεφάλαιο που αφορά την προστασία, μιλάει για την απόφαση ε, του 2008 του Συμβουλίου, όμως ήδη είχαμε τα, ε, την απόφαση, τη, συγγνώμη, την οδηγία για τα αστυνομικά δεδομένα Έχουμε μία νέα οδηγία προστασία δεδομένων για τα αστυνομικά δεδομένα με μία δικλίδα ασφαλεία ε, ε, επικαιροποιημένη. Πότε θα επικαιροποιηθεί και ε, η απόφαση Συμβουλίου ΠΡΟΥΜ για καλύτερη παροχή προστασία που θα συνάδει με του νέου κανόνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ένστ νομίζω έφυγε εντωμεταξύ. Η FTD δεν είναι εδώ. Η ND δεν είναι εδώ. Οπότε περνώ στους ευρωβουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κίνγκ που παρίσταται εδώ σήμερα και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητά του για τα θέματα που μας παρουσίασε, αλλά είπατε και εσείς ο ίδιος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και μάλιστα είναι εξόχως σημαντικά δεδομένων των κινδύνων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μιλάω μόνο για το ΠΡΟΥΜ, αλλά μιλάω και για το PNR. Δεν ε, υπάρχει ακόμη πλήρης εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Σας ερωτώ λοιπόν, ποιες είναι οι δυσκολίες. Είναι καθαρά οικονομικής φύσεως, χρηματοδοτικής φύσεως ε, και για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διαφορές, γιατί δεν προβλέψαμε ένα, μια οικονομική στήριξη. Ήταν επαρκής η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Μιλήσατε επίσης και για παρακολούθηση. Πολύ χρήσιμο μου φαίνεται αυτό για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη τα υπόλοιπα, τα 13 που απομένουν, για να μπορέσουν να μεταγράψουν την οδηγία PNR στην νομοθεσία τους. Μας μιλήσατε για παράδειγμα για ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, εν προκειμένου. Μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία PNR. Και ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο έθεσαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, το θέμα της ασφάλειας των δημοσίων χώρων και των ε, σημαντικών ε, ε, υποδομών. Μιλάμε για την ασφάλεια των μεταφορών και συζητούμε στην Επιτροπή για την Τρομοκρατία αυτό το θέμα, αλλά Υπάρχουν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, υπάρχουν τα λιμάνια. Όλε οι υποδομέ που αφορούν τη μεταφορά είναι πολύ σημαντικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει μελετήσει αυτό το θέμα. Περιμένουμε, θα μπορούμε να, μπορούσαμε να περιμένουμε μία επέκταση της οδηγίας και σε αυτό το θέμα, ο κύριος Λένερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Κίνγκ, για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Είπατε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά την ασφάλεια. Συμφωνώ και σας ευχαριστώ για όλες τις πρωτοβουλίε που έχετε αναλάβει ω τώρα και μου κάνει εντύπωση να ακούω του συναδέλφου να λένε ή να αμφισβητούν κατά πόσο πρέπει να κάνουμε περισσότερα στον τομέα τη ε, ασφάλεια, γιατί ε, οι εγκληματικέ στατιστικές πέφτουν, ε, πέφτουν συνεχώς. Είναι σαν να λέμε ότι εφόσον πέφτει η ανεργία δεν πρέπει να προσπαθούμε να ενισχύουμε την απασχόληση. Πράγματι, συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τι προκλήσει ασφάλεια για το μέλλον και νομίζω ότι παίζει βασικό ρόλο το PNR σε αυτό. Λίγο με απογοητεύει το ποσοστό εφαρμογή οδηγία PNR. Πολλά χρόνια εργαζόμαστε επί αυτού του ζητήματο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά είχε κατηγορηθεί και ω ΕΛΚ εμεί συμφωνούσαμε ότι λιγάκι καθυστερούσαμε ως προς αυτό το θέμα και τελικά καταφέραμε να υπάρχει μια συμφωνία και εγώ θα περίμενα όλα τα μέλη του Συμβουλίου, όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν μια προσπάθεια εφαρμογής και ε, είμαι κάπως απογοητευμένος. Υπάρχει έλλειψη μεταγραφής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και αυτό επηρεάζει βέβαια το σύνολο της εφαρμογής του PNR όπως είπατε κι εσείς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν ε, έχω μία ερώτηση που συνεχίζει αυτό που ρώτησε η κυρία Γκρίσπεκ ε, τι ε, ενδοενωσιακές πτήσει μεταξύ των κρατών μέλων της Ένωσης. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτά. Αν η έλλειψη μεταγραφής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη επηρεάζει την εφαρμογή του PNR, πώς η έλλειψη της γενικής εφαρμογής, ομοιόμορφης εφαρμογής, ε, τότε ε, πώ επηρεάζεται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του PNR στο σύνολό του. Ευχαριστώ πολύ. Γκόμε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, εγώ από την αρχή, εγώ ρωτώ τι κάνουν τα κράτη-μέλη όταν έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα κενά που υπάρχουν στο PNR ε, όσον αφορά τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τις charter πτήσεις και τα μικρά αεροδρόμια. Αλλά θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Αν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια, για την αντιμετώπιση όλων αυτών των κενών, αν εγώ ήμουν μαχητής στη Συρία και ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ευρώπη, εγώ θα πήγα στη Λιβύη, θα ερχόμουν σε επαφή με την με τις παραστορικές οργανώσεις στο Τρίπολη. Θα, ε, θα καλούσα τον, ε, τον ε, υπεύθυνο στη Μάλτα για να πληρώσω μια χορήγηση θεώρησης. Τρία χιλιάρικα θα έδινα. Το 2013-2014 έδωσε περίπου 88.000 ε, θεωρήσεις. Πάω λοιπόν στη Μάλπα και μετά παίρνω ένα φέρι, το είδαμε και στην Κατάνια, ένα, το, αυτό το τεράστιο φέρι, ε, ε, με, με νιολογημένο στη μαλέτα, ε, έχω και το συγκεκριμένο αριθμό, έχω και τις φωτογραφίες ε, και είμαι στην Κατάνια, στην Ιταλία. Έχω φτάσει. Πολύ εύκολο, πανεύκολο. Κάθε μέρα μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ έγραψα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και πολλά, πολλοί άλλοι συνάδελφοι για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τι γίνεται λοιπόν, διερευνάται αυτή η υπόθεση. Επίση, ένα αστυνομικό στη Μάλτα που ήταν αυτό που ε, διαχειριζόταν ε, τέλο πάντων αυτέ τι θεωρήσει. Ε, συνελήφθη γιατί είχε αποσπαστεί στο αεροδρόμιο και δεν επέτρεπε σε όσου δεν είχαν θεωρήσει να περάσουν στη ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο? Όχι? Εντάξει. Τότε θα ήθελα κι εγώ να κάνω μερικέ ερωτήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέμα του αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα ή λιγότερα είναι σημαντικό. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Δεν είναι απλώ ένα τεράστιο θέατρο ασφάλεια. Γιατί τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. είναι σαν τις κινέζικες μαριονέτες. συστηματικά δεν υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου για καμία πρόταση που αφορά την ασφάλεια. Αυτό είναι συστηματικό. Ποτέ δεν γίνονται τέτοιε μελέτε ε, και σε, καμία άλλη, σε κανένα άλλο τομέα δεν θα ήταν αυτό αποδεκτό. Δεύτερον, Υπάρχει λίγη ή σχεδόν καθόλου εφαρμογή. Δεν είναι μόνο το PNR και το PRIM. Θυμάστε την ε, κράτηση των ε, δεδομένων, την αποθήκευση των δεδομένων. Ε, ε, το είχαμε πει, αλλά πολύ λίγα κράτη-μέλη το εφήρμοζαν. Ένα συνταγματικό δικαστήριο στο ένα ή στο άλλο κράτο μέλο για κάποιο λόγο το σταματούσε. Το θέμα των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των διαβατηρίων. Μάθαμε τώρα ότι 7 χώρε, 7 χώρα, 7 χώρες συμπεριλαμβανομένη Ελβετίας ανταλλάσσουν δεδομένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να σας αποκαλύψει. Γερμανία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία και Αλβετία. Εγώ σας τα αποκαλύπτω. Αυτά είναι τα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ υπάρχει μία νέα πρόταση επιτάπητος για δακτυλικά αποτυπώματα στις αστυνομικές ταυτότητες. Και εγώ αναρωτιέμαι, όπως κάνει και ο κύριος Λίναρντ, ε, θυμάμαι όταν οι συνάδελφοί σας στο ΕΛΚ μας είπαν, όταν εγώ δεν ήθελα να... Ε, κάνουμε νωρίτερα την ψηφοφορία, είπατε ότι η επόμενη επίθεση θα πέσει στο δικό σας το κεφάλι. Εσείς θα φθέτε. Το κρίμα θα είναι στο λαιμό σας. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι 10, 15, 17 κράτη-μέλη. Εγώ θέλω να καταλάβω τι είναι πίσω από αυτό. Για ποιο λόγο μας λένε ότι πρέπει να υπογράψουμε και όταν κάνουμε ερωτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα μας λέτε ότι καθυστερούμε. Ότι καθυστερούμε πίτιδες. Γιατί για το PNR μπορώ να σας πω ότι δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο παραγνωρίζεται παντελώς από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν να μην υπάρχει, αλλά και στη δική μου χώρα, δεν λέω τίποτα για την κυβέρνηση, γιατί η δική μου θέση είναι σαφής ως προς αυτό, το ανώτατο νομικό σώμα στην Ολλανδία λέει ότι έτσι όπως είναι τώρα ε, η νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως είχε γίνει και με την αποθήκηση των ε, δεδομένων και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Όμως εξακολουθεί να πιέζει, εξακολουθούν να πιέζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατη σε αντίθεση με ε, όλους τους διακανονισμούς. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για τα αστυνομικά, για την αστυνομική συνεργασία, τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το επιθυμούσαν αυτό. Ε, και υποθέτω ότι εφόσον τους ενδιέφερε τόσο πολύ, μέχρι τις 6 Μαΐου ε, θα είχαν περισσότερα κράτη-μέλη θα είχαν εφαρμόσει. Δύο τα εφάρμοσαν μόνο και τώρα υπάρχουν 26 διαδικασίες επί παραβάζει για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν το εφαρμόζουν. Εν ολίγης, Όλοι λένε, συνεχώ το ακούω αυτό, ότι είναι σημαντικό, είναι χρήσιμο, είναι κεφαλαιόδου σημασία για την αντιμετώπιση του εγκλήματο. Δεν ξέρουμε όμω, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί δεν υπήρξε μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου, δεν υπήρξε αξιολόγηση. Εδώ η έκθεση δείχνει ότι οι στατιστικέ ε, που υποστηρίζουν τις σχετικές, ε, τους σχετικούς δεν υφίστανται. Μπορεί να υπάρχουν οι και να ισχύουν. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για το κατά πόσο θέλουμε περισσότερα ή λιγότερα, εγώ θα ήθελα να πω, θα ήθελα να μάθω τι έχουμε αυτή τη στιγμή, τι εμποδίζει τα κράτη-μέλη από την εφαρμογή, πόσα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξοδεύονται και τι κρατάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίσω από το να πιέσει τα κράτη-μέλη να, εφαρμογή, να, να περάσουν στην εφαρμογή. Εγώ δεν είμαι έτοιμη να ψηφίσω κανένα άλλο νομοθέτημα πριν καταλάβω για ποιο λόγο ε, μας ε, το φέρνουν καπέλο ε, και μας υποχρεώνουν ε, να το εφαρμόσουμε. Εφτά χρόνια το συζητάμε αυτό. Είπατε 17 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει το PNR, 20 όμως θέλουν να εισαγάγουν και τις ενδοενωσιακές πτήσεις ε, θέλουν λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τις πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν το καταλαβαίνω. Ε, τι να σας πω. Αν εγώ δεν καταλαβαίνω, κατηγορήστε με ότι δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω πως όλα αυτά φέρνουν περισσότερη ασφάλεια. Έχετε όσο χρόνο θέλετε να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς, δεν ακούμε. Uh, um, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κάποιος είπε ότι διαθέτω αίσθηση του χιούμορ. Βοηθάει επί του παρόντος. Το ζήτημα που συζητάμε σήμερα όμως είναι σοβαρό και προσωπικά το παίρνω πολύ στα σοβαρά όλη αυτή την συζήτηση, τις λεπτομερείς ερωτήσεις που κάνατε, αλλά και την αγανάκτηση που, που διακρίνω σχετικά με το πώς προχωράει η, η δουλειά μας σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι δικός μου τομέας να πω αν χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη ασφάλεια τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζοντας τις προτάσεις μπορούν να μας δώσουν και το δικό τους feedback πάνω στο ζήτημα αυτό. Δεν θα επισέλθω επομένως σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση που δεν πιστεύω ότι θα ήταν παραγωγική σχετικά με περισσότερη ή λιγότερη ασφάλεια. Προσωπικά πιστεύω ότι οποιαδήποτε επίθεση και πιο συγκεκριμένα τρομοκρατική επίθεση είναι μια συνολική επίθεση και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην υπάρχει περιθώριο τέτοιων επιθέσεων. Θέλω όμως να επιστρέψω σε ένα-δύο σημεία που θίξατε. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την φύση της προσέγγισής μας. Δεν πιστεύω ότι ποτέ χρησιμοποίησα γλώσσα του τύπου η επόμενη επίθεση θα είναι δική σας ευθύνη, σας φοράω καπέλο τη μία την άλλη απόφαση ή ότι σας κατηγορώ προσωπικά να καθυστερείτε επίτηδες. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησα ποτέ τέτοιες εκφράσεις και αν ποτέ το χρησιμοποίησα απολογούμε, υποδείξτε μου πότε το είπα και θα ζητήσω συγγνώμη. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, λέει ο Επίτροπος, και μετά θα πάρετε το λόγο στην Πρόεδρο. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ποτέ μίλησα κατά αυτόν τον τρόπο τα τελευταία χρόνια που εργαζόμαστε. Αν όμως πιστεύετε ότι το έκανα, παρακαλώ υποδείξτε μου πότε και θα απολογηθώ. Αυτό που παίρνω πολύ στα σοβαρά είναι ότι η προσέγγιση μας στον τομέα αυτό προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ριζωμένη σε αξιολογήσεις αλλά και σε γεγονότα. Συμφωνώ 100% ότι αν ξεκινάμε κάτι είναι ανάγκη να εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε. Και αν δεν το κάνουμε, τότε δεν μπορούμε να είμαστε επιτυχείς, αλλά δημιουργούνται και αμφιβολίες για περαιτέρω προτάσεις. Συμφωνώ, το δέχομαι αυτό. Πάντοτε το δεχόμουν. Αυτό που δεν δέχομαι είναι ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση κάθε μεμονωμένης πρότασης. Σε, αυτά που είπατε λοιπόν, εγώ έχω να αντιτάξω 15 χρόνια ενδελεχών αξιολογήσεων, τις οποίες και σας τις παρουσίασα. Δεν με ρωτήσατε ποτέ κάτι για τις αξιολογήσεις αυτές. Σας έδωσα το έγγραφο αυτό. Ήρθα σε εσά και σας είπα μπορούμε να έχουμε μια λεπτομερή συζήτηση και δεν υπήρξε συζήτηση, απλά προχωρήσαμε. Δεν είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν κάνουμε μελέτες αντικτύπου. Ίσως να ίσχυε πριν την, τον, την δική μου έλευση. Αποδέχομαι την κριτική αυτή εξ αρχής την αποδέχτηκα. Έχουμε κάνει όμως μελέτες αντικτύπου στις πρόσφατες προτάσεις μας. Μπορεί να μην σας αρέσουν τα αποτελέσματα, μπορεί να μην θεωρείτε ότι είναι όσο ενδελεχείς θα έπρεπε, ωστόσο έχουν γίνει μελέτες αντικτύπου. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου για τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, για παράδειγμα. Και αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα της δικής μου δέσμευσης, το οποίο και σας έχω ανακοινώσει ε, σε ό,τι αφορά την δέσμευσή μου για να βασίσουμε σε γεγονότα τη χάραξη πολιτική σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντική και είμαι εξίσου αγανακτισμένο, σα διαβεβαιώ, ο καθένα από εσά εδώ. Γιατί δεν τα πάμε όσο καλά θα έπρεπε σε ορισμένους τομείς ό,τι αφορά την εφαρμογή. Κυρίως σε, αυτά, σε αυτές τις υποθέσεις που τραβάνε πολύ σε μάκρος, για παράδειγμα το PNR. Δεν είναι ε, προς άμυνά μας να σας λέω ότι τα πάμε καλά κάπου και κάπου αλλού. Όχι. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε Uh, σε ό,τι αφορά την οδηγία δεν ε, βρισκόμαστε στο επίπεδο που θα ήθελα. Έχουμε μέχρι στιγμής μόλις εννέα μέλη που έχουν ε, περάσει σε μεταγραφή νομοθεσίας της συγκεκριμένης οδηγίας και θέλω να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο της οδηγίας αυτής όσο πιο ενδελεχώς γίνεται. Σας παρακαλώ λοιπόν να δυσκολέψετε τη, τη δουλειά μου στους τομείς αυτού, σε όλους τους τομείς. Η κριτική σας με ενδυναμώνει ούτω ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε περαιτέρω τα, τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή όλων αυτών των οδηγιών. Σε ό,τι αφορά το PNR, είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Μέχρι στιγμής έχουμε 15 που επισήμως ε, μας έχουν ενημερώσει για τη μεταγραφή της νομοθεσίας. Έχουμε 27, είναι μόλις 27 τα μέλη ο στόχος μας. Μας έχουν στείλει μια λίστα των αρμόδιων αρχών που μπορούν να λαμβάνουν PNR στοιχεία και να τα επεξεργάζονται. 22 από τα 27 μέλη έχουν ενημερώσει τις διάφορες μονάδες. 24 μέλη μας έχουν ενημερώσει για την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν την νομοθεσία σε πτήσει στο εσωτερικό της Ένωσης. Για να απαντήσω όμως την ερώτησή σας, μέχρι ότου έχουμε όλα τα στοιχεία της εφαρμογής, δεν μπορούμε να, να είμαστε σίγουροι. Ωστόσο, αυτά τα, αυτά τα νούμερα που σας είπα τώρα δείχνουν κάποιο πρόοδο. Μπορεί να μην είναι επαρκή. Και εσείς θα πρέπει λοιπόν να, να πιέζετε μένα για να πιέζω εγώ τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την αστυνομία έχουμε 8 κράτη-μέλη. Κάποιοι έχουν ε, θίξει το ζήτημα, αλλά όχι όσο πρέπει. Και πάλι, λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι εδώ μπροστά σας ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών αυτών. Τώρα σε ό,τι αφορά τις πιο λεπτομερείς ερωτήσεις σας. Το ερώτημα των υποθέσεων PNR. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό ερώτημα. Αν ισχυριζόμαστε το PNR χρησιμοποιείται και για την επιβολή του νόμου και όχι μόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έχουμε θετικό feedback με συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα παραδείγματα από τα κράτη-μέλη. Ρωτάτε γιατί δεν ε, λέμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό εδώ το πλαίσιο. Αν ε, είχαμε μια συνάντηση όπου θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε πιο ευαίσθητες πληροφορίες, πιο απόρριτες πληροφορίες, θα μπορούσαμε να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν μιλάω με τα κράτη-μέλη, μου δίνουν, έχω στη διάθεσή μου πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Την προηγούμενη φορά που ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είδα ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα μπροστά στα μάτια μου να εκτιλήσετε. Κάποιος εγκληματίας α, τον σταματήσανε μπροστά στα μάτια μου με βάση τα δεδομένα αυτά. Ε, είναι χαρά μου να μοιραστώ τέτοιου τύπου παραδείγματα μαζί σας. Όχι όμως αυτό εδώ το περιβάλλον. σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ανταλλαγής δεδομένων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, προσωπικά στηρίζω την ενδυνάμωση αυτής της υποχρέωσης ανταλλαγής δεδομένων. Έχουμε συμφωνήσει σε συγκεκριμένα βήματα ούτω ώστε να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη να ανταλλάζουν δεδομένα σε αφορά την τρομοκρατία. Είμαι απολύτως ανοιχτό σε αυτή την προοπτική. Υπάρχει μία πρόκληση σε ό,τι αφορά το PNR. γιατί θέλουμε η ανταλλαγή δεδομένων να είναι όσο το δυνατόν πιο εκτενής, όταν συμφωνήσαμε ε, για την οδηγία PNR, δεν είχαμε προβλέψει την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων. Υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη εξισορρόπησης ανταλλαγής δεδομένων με πάρα πολύ πληροφορία. Και αυτό που αποφασίσαμε τότε ήταν ότι τα κράτη-μέλη μέσω των δικών τους μονάδων θα πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν κάπως τα αποτελέσματα, τα δεδομένα. Διαφορετικά θα ήταν άχρηστα τα δεδομένα. Είπαμε λοιπόν ότι τα απαραίτητα στοιχεία α, ε, υπησερχόταν το στοιχείο της κρίσης από το κάθε κράτος μέλος. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε λεπτομερώς είναι πώς τα πάει αυτή η ανταλλαγή δεδομένων στην πράξη. Αν γίνεται ανταλλαγή σχετικών χρήσιμων δεδομένων, είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε ευχαριστημένοι ή πρέπει να το επανεξετάσουμε. Έχοντας πάντοτε κατά νου την ισορροπία μεταξύ χρήσιμων στοιχείων, ανταλλαγή στοιχείων και να μην πνιγούμε στις πληροφορίες. Αυτό είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ σχετικό ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τα κενά τώρα στο PNR. Ένα ζήτημα που έχουμε θίξει και προηγουμένως. Και η κυρία Γκομές ε, κάνει καλά και μας αγκαλεί σε αυτό το, το ζήτημα. Δεν είναι μόνο οι πτήσεις τσάρτερ. Είναι και η χρήση άλλων αεροπλάνων που πραγματικά πετάνε εκτός συστήματος. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Ίσως πιο σαφής από ότι ήμουν σε, προηγούμενους, σε προηγούμενες συζητήσεις. Να, να προωθήσουμε το διάλογο αυτό. Αναγνωρίζω ότι δεν απαντά σε όλα σας τα ερωτήματα, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε οντότητες και άτομα που χρησιμοποιούν αεροπλάνα για εμπορικούς σκοπούς και άτομα που χρησιμοποιούν αεροπλάνα για μη εμπορικούς σκοπούς. Επομένως, αν είστε μια οντότητα, μια επιχείρηση, ένα άτομο που χρησιμοποιεί, δανείζει, με συγχωρείτε, το ή τα αεροσκάφη της σε όλους, μόνο για να πετάξουν, τότε πιστεύουμε ότι αυτό υπόκειται στην κατηγορία των γενικών πτήσεων, σύμφωνα με την οδηγία PNR. Επομένως, οι πτήσεις charter θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην οδηγία PNR. Θέλω να είμαι σαφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε. Αποκινούμε τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του PNR πάντα. Η εφαρμογή του PNR αφήνει λίγο περιθώριο σε μικρές αεροπορικές εταιρείε. Η γραφειοκρατία είναι λίγο πιο εύκολη για αυτούς. Παρ' αυτά δεν εξαιρούνται όμως από την οδηγία. Οι πληροφορίες που ανταλλάζουν, που μοιράζονται μπορεί να μοιάζουν περισσότερο με ένα έγγραφο Word ή με ένα έγγραφο Excel, μπορεί να είναι και απλά email, ηλεκτρονικά μηνύματα. Δηλαδή είναι λιγότερο λεπτομερής από τις πληροφορίες που παίρνουμε από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύουμε ότι θεωρούμε ότι υπόκεινται στην οδηγία PNR αυτού του τύπου η ανταλλαγή πληροφοριών. Και αυτό είναι α, κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε και με τα κράτη-μέλη. Δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις της κυρίας Γκόμες αλλά πιστεύω ότι μπορούμε λίγο να, από κοινού να κλείσουμε κάποιες τρύπε. Για τις διαφορές μεταξύ του ε, ενδοενωσιακού και του διεθνούς PNR. Ξέρω ότι σας ε, απογοητεύει πολύ η κατάσταση και εμένα με απογοητεύει. Στο διεθνές PNR πρέπει να προχωράμε σταδιακά βήμα το βήμα Υπάρχει εντολή για τις συζητήσεις με τους Καναδούς. Κάναμε τον πρώτο γύρο συζητήσεων, όπου συζητήσαμε και για το πώς θα σεβαστούν την απόφαση του δικαστηρίου στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Σαρτζεντίνη. Στο παρελθόν υπήρξε παράδοση που θέλω να σεβαστώ ότι όσο προχωρούν αυτές οι διαπραγματεύσεις ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο. Ε, παραλαμβάνω ότι δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει στο παρόν πλαίσιο, αλλά αν βρούμε ένα άλλο πλαίσιο που έχουμε αξιοποιήσει και στο παρελθόν, τότε δεσμεύομαι να σταλεί κάποιο και να σε ενημερώνει τακτικά ή και εγώ ίδιος εάν συμμετέχω προσωπικά στις ε, διαπραγματεύσεις για το πώς πάνε. Γιατί θέλουμε να υπάρξει πλήρης ε, διαφάνεια εναντίμων. Τώρα, θα συνεχίσουμε να προχωράμε την εφαρμογή της οδηγίας για το νοσιακό PNR. Αν ε, πρέπει να ξαναδούμε λόγω της απόφασης του δικαστηρίου ορισμένα στοιχεία ε, αυτού του εσωτερικού PNR θα το κάνουμε. Αλλά και εσείς ε, και εμείς αναγνωρίζουμε ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Η απόφαση του δικαστηρίου για τον Καναδά είχαν να κάνουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός νομικού μέσου, δηλαδή μιας διεθνούς συμφωνίας που επιτρέπει σε μια τρίτη χώρα να συλλέξει στοιχεία για τους πολίτες της Ένωσης που μεταβαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα. Αυτή είναι η βάση της απόφασης του δικαστηρίου για τον Καναδά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη υπάρχει κάποια αναλογία για το ενωσιακό PNR όπου η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Είναι για λόγους επιβολής του νόμου, κατά πολέμης, τρομοκρατίας, όχι για ελέγχους στα σύνορα ή για έλεγχο της μετανάστευσης. Και ιδιαίτερα για τις ενδοκινητικές πτήσεις. Δεν, δεν βγαίνουν από την ε, επικράτεια της Ένωσης. Άρα πρέπει να δούμε τι στοιχεία αυτής της απόφασης αφορούν το εσωτερικό PNR και θα το κάνουμε. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις για το PNR. Α, όχι, όχι, όχι. Και η επέκταση του PNR σε άλλες μορφές μεταφορών και μετακίνησης. Η οδηγία του PNR δεν δίνει εντολή στα κράτη-μέλη να το διευρύνουν σε άλλες μορφές μεταφορών, αλλά ούτε το αποκλείει και γίνονται συζητήσεις μεταξύ κάποιων κρατών μελών μεταξύ τους για παράδειγμα για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να μας απασχολήσουν για λόγους ασφαλείας ιδιαίτερα γιατί έχουν υπάρξει επιθέσεις σε σταθμούς άρα έχει να κάνει με την προστασία των δημοσίων χώρων και σε τρένα Γι' αυτό μόλις δημοσιεύσαμε τον περασμένο μήνα ένα αναλυτικό πρόγραμμα δράσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων όπου καλύπτουμε πολλά θέματα για τη χρήση των σιδηροδρομικών μεταφορών από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και λέμε ότι η χρήση του PNR συνδέεται με αυτή μας τη δράση, με αυτό το πρόγραμμα δράσης. Αυτές είναι οι ερωτήσεις για το PNR τώρα. Τώρα, για το πριν... Λοιπόν, να απαντήσω σε μία λεπτομεριακή ερώτηση για την επίπτωση του πριμ στις τελευταίες, τι μάλλον, τις επιπτώσεις επί του πριμ των τελευταίων αλλαγών στην προστασία δεδομένων. Βεβαίω και το πριμ περιέχει μέτρα για την προστασία των δεδομένων που πρέπει να σεβαστούν τα κράτη-μέλη και ελπίζω να τη σέβονται. Σωστό είναι, όπως είπε η κυρία Σαρτζεντίνη, αν το κατάλαβα καλά, ότι η οδηγία για τις αστυνομικές αρχές λέει ότι μέχρι τις 6 Μαΐου του 19 η Επιτροπή θα επανεξετάσει και άλλα νομοθετικά μέτρα της Ένωσης που πρέπει κτλ. κτλ με στόχο να τις ευθυγραμμίσει με αυτήν την οδηγία και να γίνουν αυτές οι προτάσεις για να, που χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτή η ευθυγράμμιση. Θα συμμορφωθούμε με αυτή την ε, διάταξη. Θα επανεξετάσουμε και θα ενημερώσουμε το δίκτυο ΠΡΙΜ ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι συμμορφούνται με τις αλλαγέ στο πλαίσιο τη προστασία δεδομένων. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό. Γιατί καλούμε τα κράτη-μέλη να κάνουν πράγματα που μέχρι τώρα δεν έκαναν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνουν αυτά, τώρα θα πρέπει να γίνουν. Βεβαίω, δεσμεύομαι ότι θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ακόμη και αυτά τα θέματα που τα έχουμε τόσα χρόνια μπροστά μα. και μέσω κοινοτικών πόρων που θα δαπανηθούν προς τα κράτη-μέλη. Οι πόροι που έχουν δαπανωθεί για το ΠΡΙΜ ε, χαιρετίστηκαν από ορισμένου, από άλλους όχι. Επίσης και για το PNR ε, δαπανούμε πόρου που ορισμένοι θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να δαπανούνται και άλλοι όχι, αλλά εν πάση θα ελέγξουμε και τα κράτη-μέλη για το αν αξιοποιούν ε, τους κοινοτικούς πόρους. Και όπου είναι αναγκαίο, θα ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση. Υπάρχουν ήδη για το ΠΡΙΜ ε, πολλές τέτοιες διαδικασίες επί παραβάση. Διάφορα κράτη-μέλη ε, ξύπνησαν μετά την τις διαδικασίες αυτές και συμμορφώθηκαν, τέσσερα όμως όχι. Και για το PNR, ήδη αυτό το μήνα ξεκινάμε, θα στείλουμε επιστολές για τις χώρες που καθυστερούν. Με πλήρη διαφάνεια. Θα σας ενημερώσουμε πώς πάνε τα θέματα αυτά με αυτές τις χώρες και το πώς τις ελέγχουμε. Και μία τελευταία ερώτηση. Α, όχι, όχι. Δύο τελευταίες ερωτήσει. Πρώτον, μία που νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω καλά και μία που δεν είμαι τόσο σίγουρο. Θα έρθει ο κύριο Αβραμόπουλος αργότερα. Α, όχι. Καλά. Αν χρειαστεί θα σας γράψω κιόλας, θα σας στείλω μια επιστολή, γιατί θεωρώ ότι οι πωλήσει προξενικών θεωρήσεων και με έχετε ρωτήσει και στο παρελθόν για τις πωλήσει ηθαγένειας. Μας ανησυχούν όλα αυτά και θα πρέπει να τα εξετάσουμε από πλευράς ασφαλείας. Συμφωνώ. Τώρα τι συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής μπορούν να ληφθούν. Δεν είναι τόσο προφανές. Το συζητάω με τον κύριο Αβραμόπουλο και άλλους και αν μπορέσω να καταλήξω σε καλύτερη απάντηση αργότερα θα το κάνω, εφόσον δεν θα μιλήσετε με τον Δημήτρη. Και τέλος, για την παραπληροφόρηση. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση, κυρία Ζήπελ. Είναι κάτι που είναι πραγματικά στο επίκεντρο της δουλειάς μας για την ασφάλεια. Ιδιαίτερα εν ώψη και των ε, επικείμενων ευρωεκλογών. Δεν έχουμε ακόμη στοιχείο ότι κάποιο θα επιχειρήσει να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία. Αλλά αν δούμε τι έχει γίνει σε πρόσφατες εκλογές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, είναι πραγματικά αναγκαίο προληπτικά από την πλευρά μας να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο παρέμβασης και επηρεασμού των ευρωεκλογών σε όλες τις χώρες της Ένωσης ε, την επόμενη άνοιξη. Γι' αυτό έχουμε δύο κατευθύνσει. Μία έχει να κάνει με την ασφάλεια των εκλογών. Έχουμε κάνει μια σειρά συναντήσει. Η κυρία Γιουρόβα και εγώ και ο Φραντς Τίμερμαν. Θα έχουμε μια σειρά από συναντήσει μέχρι τον Νοέμβριο όπου θα συζητήσουμε με ανθρώπου που οργανώνουν εκλογέ και με εμπειρογνώμονε για κυβερνοασφάλεια, για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Είναι βεβαίω ευθύνη των κρατών μελών η διεξαγωγή των εκλογών αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να εξοπλίσουμε τους οργανωτές των εκλογών παντού στην Ένωση για να πάρουν τάχιστα τα αναγκαία βήματα για να δυσχεράνουν οποιαδήποτε επίθεση κατά της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, είναι ένα ευρύτερο θέμα που έχει να κάνει με την παρέμβαση εκλογές. Οπότε μια άλλη κατεύθυνση της εργασίας μας είναι η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Μαζί με την Μαρία Γαβριέλ αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε έναν κώδικα δεοντολογίας με τις μεγάλες ε, επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους φορείς για να αυξηθεί η διαφάνεια, η εχνηλασιμότητα και η λογοδοσία για τη χρήση του ίντερνετ. Ιδιαίτερα για τις ενημερώσεις του ίντερνετ, τα λεγόμενα news ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους ε, πολίτες να είναι ε, ενημερωμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν παρεμβαίνουμε ε, στο εάν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει, αλλά θα πρέπει να γίνει ευχερέστερο, να διαπιστώσουμε, για παράδειγμα, αν κάποιος είναι πίσω από κάποια προφορία, εάν κάποια προφορία προέρχεται από bot και όχι από ανθρώπους, και κάτι άλλο που συζητάμε τις μεγάλες πλατφόρμες στο ίντερνετ, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι χρήστες να ρωτάνε περισσότερο τα news feed που ε, διαβάζουν. Είδαμε ότι κάποια τέτοια θέματα τα συζητάμε με το Facebook, όπου σημειώνεται πρόοδος, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είπαμε ότι αρχικά θα είναι σε θελούσια βάση, αλλά είπαμε και δημοσίως ότι είναι επαρκώς σημαντικό το θέμα αυτό, οπότε αν δεν υπάρξει επαρκής πρόοδος ε, μέσω εθελούσιας ε, δέσμευσης, τότε θα εξετάσουμε και άλλα μέτρα για να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να καταπολεμήσουμε την παραπροφόρηση. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν κάλυψα κάποια σημεία, με χαρά να σας απαντήσω γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ζίπελ ζήτησε το λόγο για να δευτερολογήσει. Ε, ναι, ευχαριστώ. Επίτροπε King, θέλω να σας μιλήσω γερμανικά. Ορισμένα τμήματα της ομιλίας σας μου έδωσαν την εντύπωση ότι ήταν όλα θαυμάσια μέχρι τώρα. Αλλά δεν δώσατε συγκεκριμένες απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα. Και η κατεύθυνση των απαντήσεων δεν βοηθάει. Είπατε πως δεν είναι δικό σας καθήκον να αποφασίσετε αν χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη ασφάλεια. Νομίζω πως είναι επικίνδυνη αυτή η διατύπωση. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα μετάφρασης. Το θέμα δεν είναι λιγότερη ή περισσότερη ασφάλεια. Το θέμα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Οι πολίτες μας πρέπει να προστατεύονται από την τρομοκρατία και την, ε, και την εγκληματικότητα. Εάν για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα, ή ε, ισχύουν τα ίδια αποφασιστέντα. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Και πολλές εκθέσεις που έχω από διάφορα κράτη-μέλη μου λένε ότι σε πολλά κράτη-μέλη, δηλαδή εξάρτητα από το βαθμό εφαρμογής, είναι ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν έχει καμία συγκεκριμένη επίπτωση η εφαρμογή. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός των αρχών, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, μπορώ να το πω και στη Γερμανία. Πολλοί υπάλληλοι, για παράδειγμα, στην Γερμανία, πολλοί αστυνομικοί υπάλληλοι, κάνουν τρομερέ υπερορίε. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να θέσουμε. <clears throat> για το θέμα του PNR, είπατε πω δεν μπορείτε να δώσετε σε αυτό το πλαίσιο συγκεκριμένη πληροφόρηση. Μα δεν είπα να μου πείτε πώς λέγονται αυτά τα άτομα, πώς λέγεται η συμμορία τους ή πώς συνεργάζονται στο ίντερνετ. Το ερώτημά μου είναι, είναι σε αυτές τις υποθέσεις ανακαλύψαμε κάποιον που προηγουμένως δεν τον ξέραμε ή κάποιος ε, ο οποίος ε, είχαμε την υποψία ότι θέλει να κάνει κάτι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι βεβαιώνεται αυτή η καποιος ο οποιος ειχαμε την υποψια οτι θελει να κανει κατι μπορεσαμε να διαπιστωσουμε οτι επιβεβαιωνεται αυτη η υποψια και με βάση τις λειτουργίες καταλήξαμε σε κάποιες διώξεις. Νομίζω ότι είναι γενικής φύσης ε, και το πλαίσιο μας δεν δεν είναι ακατάλληλο γι' αυτό. Και για τις, ε, την παραπληροφόρηση και τις ψεύτικες ειδήσει. πρέπει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση. Πού ξεκινάει η παραπληροφόρηση, πώς την αντιμετωπίζουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Να σβήσουμε όλα όσα είναι στο ίντερνετ με το οποίο συμφωνούμε. Νομίζω ότι κατά την ε, προεκλογική εκστρατεία για το Βρετανικό δημοψήφισμα πολλά που έλεγε η Λούκε και ο, Φαρά, ο Λούκε και ο Φαράτζ ε, ήταν ψέματα. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Να το φημώσουμε. Και το θέμα στο ίντερνετ είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την παραπληροφόρηση. Τη σβήνουμε και πώς τη σβήνουμε. Δεν επιτύχαμε ακόμη την καλύτερη λύση. Χρειαζόμαστε περισσότερη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και του πολίτε μας για να μπορούν να καταλάβουν καλύτερα πώς θα αντιμετωπίσουν, πώς θα αναγνωρίσουν καλύτερα και πώς θα αμφισβητήσουν καλύτερα αυτή την παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση δεν απαντήσατε, αλλά θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι εγώ προσωπικά δεν σας κατηγόρησα εσάς προσωπικά ότι πιέσατε τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή μας, γιατί θυμάμαι αποδηλώσεις στην Ολομέλεια, θυμάμαι ανακοινωθέν που από συγκεκριμένη ομάδα ε, και ε, υπονοούσαν μια άμεση σχέση μεταξύ ε, τρομοκρατίας και συμπεριφοράς των ψηφοφόρων. Αλλά δεν το συνέδεσα αυτό με εσάς προσωπικά. Είπατε 8 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την οδηγία ε, την αστυνομική δεδομένη τη σημασία και δεδομένου του ότι πρέπει να είναι το αντίβαρο αυτή η οδηγία σε όλη αυτή τη συλλογή δεδομένων κλπ. Ε, είπατε ότι ξεκινήσατε διαδικασίες επί παραβάση για τα υπόλοιπα 22 κράτη-μέλη, γιατί είπατε ότι θέλετε να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή, αλλά δεν παίρνει κανεί βαθμούς για την προσπάθεια στο σχολείο, αλλά για τα αποτελέσματα. Αν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν ε, να εφαρμόσουν κάτι για το οποίο, ζήτησαν, το οποίο οι ίδιοι, τα ίδια, ε, τότε δεν θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερο χρόνο, δεν τους δίνεται περισσότερο χρόνο. Όχι, όχι, δεν εννοώ και εγώ ότι εσείς με κατηγορήσατε. Ε, θα ήθελα να απαντήσω στη δεύτερη ερώτησή σας με ένα κατηγορηματικό ναι. Πράγματι θα γράψουμε στα κράτη-μέλη πριν από τις καλοκαίρινέ διακοπές για όλα τα κρατη που, δεν μας, σε όλα τα κράτη-μέλη που δεν μας έχουν ενημερώσει για την εφαρμογή της αστυνομική οδηγίας. Το ίδιο πράγμα, η ίδια λογική ισχύει και γι' αυτό ε, όπως εξήγησε και στα υπόλοιπα θέματα που ε, συζητούμε. Θα του κυνηγήσουμε. Να απαντήσω στην κυρία Ζίπελ πολύ σύντομα. Υπάρχει μια συζήτηση για το σωστό επίπεδο ασφάλειας. Εγώ δεν θα το λύσω αυτό. Εμείς πρέπει από κοινού να το λύσουμε μέσω της διαδικασίας, ε, της, ε, μέσω της νομοθετικής διαδικασίας εδώ ε, και στο Συμβούλιο. Μακράνε μου να επιβάλλω κάποια ιδέα της σωστής ασφάλειας, ε, γιατί δεν θέλω να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο μιλά ο κόσμος για το σωστό επίπεδο ασφάλειας, δεν νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει. Δεν, δεν θα μπορέσουμε να επιφέρουμε την απόλυτη ασφάλεια, τη το μηδενικό κίνδυνο, αλλά φυσικά η πρόθεσή μα αυτή είναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία είναι να δούμε τομεί ο οποίο μπορούμε να λάβουμε πρακτικά μέτρα για να μειώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δράσουν όλοι αυτοί που θέλουν να μας βλάψουν, οι τρομοκράτες και οι υπόλοιποι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα ε, σε σχέση με την αντιμετώπιση των μέτρων που χρησιμοποιούνται, σε σχέση με την ενίσχυση της κρίσης των πληροφοριών που πιστεύω ότι είναι ένα βασικό ε, εργαλείο στο πλαίσιο της εργασίας αυτής και με τη σωστή προστασία που είναι κάτι το οποίο, ε, για το οποίο εσείς ε, και άλλοι ε, μου ζητάτε να είμαι αποτελεσματικός και να λογοδοτώ. Αυτή είναι μια συζήτηση που κάνουμε, αλλά αυτό το επίπεδο ασφάλειας ή το άλλο επίπεδο ασφάλειας φοβάμαι ότι ε, θα είναι μία στήρα ανταλλαγή απόψεων ε, που δεν θέλω να, ε, να συμβεί. Εγώ θέλω να μειώσω το χώρο δράσης των τρομοκρατών και άλλων όταν θέλουν να μας βλάψουν, να καταστήσω δυσκολότερη τη δυνατότητα επίθεσης και μιλάω και για τον χώρο και να μπορώ να τα αντιμετωπίσω όταν συμβαίνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα ε, στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να γίνουν συζητήσεις μα ε, Συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα. Μπορούμε να συζητήσουμε τι αξία έχουν. Ε, όσον αφορά το PNR. Κοιτάξτε. Πράγματι, βρίσκουν άνθρωπους ε, που προηγουμένως δεν τους είχαμε δει γιατί ε, βρίσκουν ε, τάσεις κάποια, κάποια πεπατημένοι που ακολουθούν οι άνθρωποι αυτοί. μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες αν θέλετε και πριν από τον επόμενο διάλογο, διάλογο για υποθέσεις που βάσει του PNR έφτασαν στη δικαιοσύνη. Να το διερευνήσω αν θέλετε. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να υπάρξει μια συνάντηση ευχαρίστω μεταξύ μα στην απαραίτητη σύνθεση ώστε να το συζητήσουμε αυτό. Όλου θα μα βοηθούσε ε, να δούμε αυτά τα πρακτικά παραδείγματα. Και τέλο, όσον αφορά την παραπληροφόρηση, και για να είμαι σαφέ και θα έχουμε και άλλες, να είμαι και θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε να το συζητήσουμε, έχουμε προτείνει έναν ορισμό. Είναι στην ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε νωρίτερα φέτος ε, είναι εσκεμμένη παραπληροφόρηση με συγκεκριμένη πρόθεση αποτελέσματος οικονομική ή πολιτική. Ε, πρέπει να λάβουμε δράση εναντίον τέτοιου είδους πληροφόρησης, αλλά δεν μιλάμε για στοχοθέτηση συγκεκριμένων, συγκεκριμένου περιεχομένου και να πρέπει κάποιος να κρίνει κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό δουλεύει. Δεν δουλεύει σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει την ανιχνευσιμότητα, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και αυτά θα επιτρέψουν ε, στα κράτη-μέλη ε, και τους χρήστες, όπως τους αποκαλεί ο κλάδος, να έχουν τη δική τους κρίση, ε, τη δική τους αξιολόγηση για αυτά που βλέπουν ή διαβάζουν. Ο τρόπος λοιπόν αντιμετώπιση της παραπληροφόρηση είναι εντελώ διαφορετικός από αυτόν ε, τον τρόπο, ε, από τον τρόπο αντιμετώπισης του παράνομου περιεχομένου. Τότε υπάρχει ένας ορισμός κοινό σε όλη την Ευρώπη, ξέρουμε γιατί μιλάμε, ε, Ξέρουμε ότι το περιεχόμενο αυτό μπορεί να εντοπιστεί και συνεπώς μπορεί κανείς να αναλάβει δράση κατά αυτού του περιεχομένου βάσει του γεγονότος ότι είναι παράνομο. Ε, δεν είναι όλα λοιπόν ε, το ίδιο πράγμα. Να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν τη διεξοδική ανταλλαγή απόψεων. Ε, νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνεται η πρωινή μας ε, συνεδρία. Δέκα λεπτά πριν ε, από την